να εξόχως από μεμακρυσμένων περιοχών. Και έχουμε επίσης και το γενικότερο θέμα της συνάντησης της διακοινοβουλευτικής με τις ομόλογες επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό θα γίνει Ελπίζω να υπάρχουν αρκετοί παρόντες, εν πάση περιπτώσει. I think EPP e is in difficult position. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι σε δύσκολη θέση γιατί δεν έχει μέλη στην αίθουσα. Μόνο το συντονιστή. Και σύν της άλλης ο Λάμπερτ δεν έχει την κάρτα του οπότε ούτε και αυτός θα ψηφίσει. So I uh, am not going to be helped. Ah, what happens here? Francis? <laughs>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

Mm. Now we can start. <laughs> Now they will discover they have no cards. Can we? <coughs> Can I just ask you? To... Λοιπόν, σας παρακαλώ να ελέγξετε αν έχετε τις σωστές κάρτες στο μηχανισμό ψηφοφορίας.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 Κοιτάξτε, η... μπορείτε να υπολογίσετε και μένα δεν είχα την κάρτα μου μαζί πάλι αυτή τη φορά. Miguel will look at Lambert all the time. So can we just start because I think okay I will start. We're starting with Luis Paulo Alves. Alves. Look. A ver, ya. Your card is not working either. Creo que I, I think my card is lost. I, I don't know whether we have... Βρίσκω την κάρτα μου. Πρόταση. Δεν ξέρω αν μπορούμε προς την Ολομέλεια. Δεν ξέρω αν ο τεχνικός μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχει τεχνικός. now it's working. Ε, yeah, but the colleagues do not have, uh, not every slot is working. So still I would like to, to suggest that if some... Λοιπόν, εάν δεν δουλεύει ε, το μηχάνημα, δοκιμάστε κάπου αλλού, δίπλα. Λοιπόν, για ηρεμήστε, γιατί είστε πολύ σήμερα έτσι δύσκολοι. Λοιπόν, για να ψηφίζουμε. Συμβαστική ένα, αλλά άλλες. Προ, Ποιος είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 σε μια άλλη σελίδα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6, επόμενη σελίδα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 Περ. κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε για λόγους που δεν γνωρίζω στην τελευταία σελίδα, στην τροπολογία 59. Στη σελίδα 7. Τροπολογία 59. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τέλειωσε. Α, τέλειο. Ψηφίζουμε λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότησης. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Μόνο ο Λάμπερτ δεν λειτουργεί, λέει η πρόεδρος. Ούτε η Ρώσα έχει την κάρτα της. Ωραία, άρα άλλοι δύο υπέρ, 35 υπέρ, 4 κατά. Μάλιστα, τελειώσαμε αυτό. So now we go to... Περνάμε τώρα στο σημείο 11, έκθεση Πακάρινεν. Οδηγία για τα καύσιμα. Τροπολογία 42, έχουμε εδώ μια προφορική τροπολογία. Είναι κάποιος κατά. Επομένως ψηφίζουμε τη 42 όπως τροποποιήθηκε. Παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε τη 42 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 20 κατά. 21 κατά. Άρα απορρίπτεται η τροπολογία αυτή. Τροπολογία 41. Ψήφι πέρα. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά μπορούμε να το ελέγξουμε. Τροπολογία 41, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Το ίδιο μου φαίνεται ότι πιο πολύ είναι κατά, αλλά στο ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 44. Υπάρχει και μια προφορική τροπολογία. Κάποιος αντίθεση με αυτήν. Όχι, άρα ψηφίζουμε. Ψήφι Κατά. Ελέγχουμε. Είναι πιο εύκολο να ελέγξουμε. Πέραση τη ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 22 προς 16. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 9 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 45 τροπολογία με προφορική. Τροπολογία είναι κάποιο αντίθετος, όχι ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, ελέγχουμε τη 45. Όπως ευτοποποιηθεί με την προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 23 ψήφι προς 16. 12 υπέρ. Κατά. Α, συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα το ελέγξουμε και αυτό. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 21 ψήφος 16 τροπολογία 46 υπέρ κατά νομίζω απορρίπτεται συμβαστική 1 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε σε τελικές σκέψεις, τα recital, τροπολογία 22 υπέρ, κατά, Ελέγχουμε την 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται 26 προς 13. Τροπολογία 1. Υπέρ. 1. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ρώσα ήσασταν κατά. Απορρίπτεται. 19 προς 20. 18 προς 20 μάλλον. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κα... Τι θέλετε. Όχι, έληξε προηγούμενη ψηφοφορία, λυπούμε. Αλλά και χωρίς τη Ρώσα ήταν, είχε απορριφθεί. 23. 23 ψήφι υπέρ. Κατά. Θα ελέγξω. 23. Πέρας. Ε, η Ρώσα και ο Λάμπερτ ψήφισαν. Υπέρ, ωραία, άρα εγκρίνεται 22 προς 18 και πηγαίνουμε στην 24 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα γρήγορα γρήγορα. Δεύτερο τμήμα τη 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα τη συμβιβαστικής 3 υπέρ. Κατά αποχέ τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Πού πάμε τώρα. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Εποχές, ναι, εγκρίνεται. Με μεγάλη διαφορά. Τροπολογή 29. Α, όχι. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Εντάξει. Τη συμβαστική 5. Δεν λέτε και στην Επιτροπή να έλθουν γιατί μάλλον θα ξεκινήσουμε νωρίτερα με το επόμενο θέμα μετά τις ψηφοφορίες. Λοιπόν, ελέγχουμε τη συμβαστική 5, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Με μεγάλη διαφορά και δεν ξέρω ποιος ήθελε να ελέγξουμε. Α, οι τέσσερις που ήταν κατά. Α, την προηγούμενη θέλατε. Α, πολύ αργά. Okay, so we go... Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήσασταν υπέρ. Κωνσταντσε τα έχασε. Λοιπόν, συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα πηγαίνουμε στην τροπολογία 33. Έχουμε προφορική τροπολογία. Είναι κάνει αντίθετο, Όχι. Ψηφίζουμε. 33. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Να ελέγξουμε την τροπολογία 6 παρακαλώ. Οι συντονιστές σήμερα δεν ξέρω, δεν τους βλέπω να τους ακολουθούν οι υπόλοιποι. Απορρίπτεται. 34 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Να ελέγξουμε όμως καλύτερα. 34. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά, νομίζω εγκρίνεται, ελέγχουμε την 35 όμως. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. 36 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά τώρα ψηφίζουμε από του συνόλου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 34 ψήφοι υπέρ, εγκρίνεται λοιπόν μεγάλη διαφορά. Και περνάμε στην οικοκαινοτομία την έκθεση του Γέννης Νίλσον. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 19 προς 20. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 7 άρχεται η ψηφοφορία λήξη εγκρίνεται τροπολογία 8 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ ελέγχουμε την 10 άρχεται η ψηφοφορία πέρασε για να ξεκαθαρίσουμε οι δύο που δεν έχουν τις κάρτες τους είναι υπέρ άρα 20 υπέρ 18 κατά άρα εγκρίνεται Νομίζω έχουμε ολοκληρώσει με τις τροπολογίες και ψηφίζουμε το σύνολο τώρα, αν συμφωνείτε. Τελική ψήφος. Ψηφίστε πιο γρήγορα παρακαλώ. Κανείς δεν θέλει να ψηφίσει. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται σχεδόν ομόφωνα. Μαρία, να συζητήσουμε τώρα το δικό σου θέμα. We have Mr. Teurer. Um, uh, dear colleagues, uh, could I just ask you for one minute attention? We... Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να περάσουμε στο 14 της Μαρία Εριγκόγεν Πέρες για την επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης. Οι συνάδελφοι που συνεργάζονται με τον Τόιρερ και τον Μαδέρη ή τον Ότζιχ, παρακαλώ ενημερώστε, μας, ενημερώστε τους ότι είμαστε εδώ. Α, ο Ότζι είναι στην Πράγα. Α, ο Γιώζιφ είναι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, η Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε ότι σε μια στην παρούσα οικονομική συγκυρία και τα μεγάλες προκλήσεις τις οποίες πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Η Ευρώπη προσπαθεί να ανακάμψει βιομηχανικά σε στρατηγικούς τομείς όπως ο αεροναυτικός τομέας, η αυτοκίνητο βιομηχανία, το διάστημα, η χημεία και η φαρμακευτική βιομηχανία είναι θα έλεγα ένα κλειδί για την αηφορία, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Ο τομέας αυτός έχει υποστεί όμως τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Έχει υπάρξει μείωση κατά 2% της παραγωγής και έχουμε χάσει 3 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Η βιομηχανία υποχωρεί και αυξάνονται φυσικά και αναπτύσσονται οι υπηρεσίες. Είναι καλές οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλουν ο τομέας αυτός να ανακάμψει. Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία επηρεάζει άμεσα τις περιοχές οι οποίες υποφέρουν από την ύφεση, από την αύξηση επίσης των ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ένωσης, στον τομέα της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής απειλείται η κοινωνική συνοχή και η εδαφική συνοχή. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια εκ νέου βιομηχάνηση της Ευρώπης μέσω αποτελεσματικών πολιτικών και κατάλληλων επαρκών οικονομικών μέσων. Είναι μία από τις βασικές πολιτικές για την ανάπτυξη της βιομηχανικής καινοτομίας, ιδιαίτερα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της σχετικές με την αηφορία την ενέργεια, της ε, κλιματολογικές αλλαγές κτλ. Για να υπάρξει αυτή η εκ νέου βιομηχάνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποια ισχυρά, τα ισχυρά ε, διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να καθοριστούν ξεκάθαρες πολιτικές βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να έχουν σαν στόχο και την κάλυψη των αναγκών στον τομέα της χρηματοδότησης, της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να απλουστευθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, να μειωθεί η φορολογία της εργασίας, να υπάρξει διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων και σε επίπεδο τοπικό και σε επίπεδο περιφερειακό και σε επίπεδο διευκόλυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γενικότερα των επιχειρήσεων. Πρέπει να ενισχύσουμε τις στρατηγικές καινοτομίες για να υπάρξει η λεγόμενη ευφυής εξειδίκευση έτσι ώστε να ακαλυφθούν οι ανάγκες από την χρηματοδότηση της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. Αυτές οι στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης βασισμένες στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιφερειών θα χρησιμοποιήσουν τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους ε, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θα πρέπει επίσης να επιδιώξουμε την βελτίωση της αποτελεσματικότητας ε, των δανείων, των εγγυήσεων και των επιδοτήσεων και όλων των μορφών οικονομικής ενίσχυσης και η σωστή λογική χρήση όλων αυτών των μέσων που θα στοχεύουν στην διευκόλυνση της διεύρυνσης στη χρηματοδότηση ανάλογα με τις ανάγκες σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνουμε και τις δημόσιες επενδύσεις και τις ιδιωτικές επενδύσεις μέσα από ένα σύστημα κρατικών επιδοτήσεων που θα δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο να καλύπτει τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Υπάρχουν και άλλες ιδέες οι οποίες θα ήθελα να συμπεριληφθούν σε αυτό το σχέδιο αλλά θα πρέπει ε, να περιοριστούμε σε ένα συγκεκριμένο αριθμό γραμμών για το μέγεθος. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σαν παράδειγμα και στην ανάγκη αύξησης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την σημασία που έχουν οι συνέργειες για την συνοχή στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής. Αλλά έχουμε προβλήματα χώρου θα έλεγα και χρόνου. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι ε, αύριο τη 12η μεσημβρινή. Στις 7 του μηνός θα υπάρξει γνωμοδότηση της ε, ήτρε και κανονικά θα πρέπει να φτάσει τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια. Περιμένω τα σχόλιά σας και τις ε, γνώμες σας τις οποίες θα συμπεριλάβω στην πρότασή μου. Ευχαριστώ. Ο είπα από πλευράς του ΕΛΚ. Και εγώ θα συμφωνήσω με την συνάδελφο κυρία Περέζ. Η εκ νέου ε, εκβιομηχάνηση της Ευρώπης παραμένει μια σημαντική πρόκληση κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης η νέα βιομηχανική στρατηγική θα είναι μια αντίδραση θα έλεγα μετά από τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη ε, και την απασχόληση στις οποίες προέβη το Συμβούλιο από το 12 και μετά. Η επιδίωξη της εκβιομηχάνησης παραμένει πάντα ένας μοχλός για την ανάπτυξη και την απασχόληση ιδιαίτερα η δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι ένας βασικός κεντρικός στόχος. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στις τεχνολογίες. Πρέπει να σκεφτούμε και το μέλλον των τεχνολογιών οι οποίες δεν θα πρέπει να επηρεαστούν αρνητικά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, τιμολόγηση του ηλεκτρισμού σαν παράδειγμα για τις βιομηχανίες γιατί τα τελευταία 8 χρόνια έχει αυξηθεί πάνω από 27%. Ε, απαιτείται μια προληπτική και προβλεπτική αντιμετώπιση θεμάτων όπως ε, οι επενδύσεις και η αηφορία. Μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιους καινοτόμους τομείς που θα οδηγήσουν στην λεγόμενη νέα βιομηχανική επανάσταση όπως οι τρισδιάστατες ε, εκτυπώσεις ή όπως τα οικολογικά φιλικά οχήματα, βιοτεχνολογίες, νανοτεχνολογίες, ε, φιλικές προς το περιβάλλον βιομηχανίες, αηφορία στην προμήθεια πρωτονυλών και αηφορία επίσης στον τομέα των μεταφορών. Να θυμίσω τον σημαντικό ρόλο τον οποίο καλούνται να παίξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι η κινητήρια δύναμη αυτής της ανάκαμψης και εμείς θα καταφέσουμε τροπολογίες στην έκθεσή σας. Δεν βλέπω κάποιον που ε, θα μιλήσει εξ ονόματος ε, της Α, ο Νίκος θα πάρει το λόγο για τους πρασίνους. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια μείωση της βιομηχανικής δραστηριότητας που οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ένα είναι σίγουρα ότι υπάρχουν, ε, ε, υπάρχει μετακίνηση βιομηχανίας εκτός των ορίων της Ευρώπης για λόγους μείωση του κόστους. Ε, υπάρχουν αλλαγές οι οποίες οφείλονται σε περιβαλλοντικές απαιτήσεις και υπάρχουν βέβαια και αλλαγές που οφείλονται στην αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών και των αξιών και των συμπεριφορών στην καθημερινή ζωή. Χρειάζεται να υπάρξει μια νέα στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, για να δημιουργηθούν και θέσει εργασία, αλλά και για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της σημερινή εποχής. Αυτή όμως η επιστροφή στη βιομηχανοποίηση στην Ευρώπη πρέπει να συνδυαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο με νέε καινοτομίε, κυρίω πράσινε οικολογικέ καινοτομίε, όπου υπάρχει δυνατότητα να συνδυάσουμε ταυτόχρονα την οικονομική δραστηριότητα με την ε, καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση των βιομηχανιών. Ε, έχουμε στήσει πολλές φορές για το θέμα της οικολογικής καινοτομία εδώ. Νομίζω ότι είναι το κλειδί απέναντι σε προβλήματα όπως είναι το ενεργειακό κόστος, ε, η αποδοχή των κοινωνιών, ε, η αποδοχή από τις κοινωνίες επενδύσεων βιομηχανικών. Όσο πιο ε, ε, υψηλή είναι η επίδοση κοινωνικά και περιβαλλοντικά των βιομηχανιών, τόσο πιο αποδεκτές μπορεί να είναι από τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί ξέρετε πλέον ότι σε πολλές περιοχές δεν είναι αποδεκτές επενδύσεις, <clears throat> επενδύσεις οι οποίες θα ρηπαίνουν το περιβάλλον και αυτό αντιμετωπίζεται εφόσον υπάρχουν πιο πράσινες επιδόσεις βιομηχανίας και πιο υπεύθυνες συμπεριφορές. Ε, καινούργια εργαλεία τα οποία έχουμε συζητήσει εδώ, όπως η βιοοικονομία, όπως είναι η γαλάζια οικονομία, είναι χρήσιμα εργαλεία για να τα συνδυάσουμε με την ε, προσπάθεια μιας νέας στρατηγικής για τη βιομηχανία στην Ευρώπη. Και σίγουρα οι επενδύσεις και η προσπάθεια αναζωγόνησης της βιομηχανίας πρέπει να συνδυάζεται με τις θέσεις εργασίας. Ε, αυτό ε, πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση ώστε η δραστηριότητα βιομηχανική να αντιμετωπίζει και τα μεγάλα προβλήματα ανεργία που υπάρχουν σήμερα. Πολλές φορές οι επενδύσεις δεν συνδυάζονται με μια τέτοια διάσταση. Είναι επενδύσεις έντασης ε, τεχνολογίας ή ένταση κεφαλαίου, αλλά πολλές φορές ο παράγοντα απασχόληση παίζει μικρό ρόλο. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much, Kelly. Θέλω να ευχαριστήσω την ισχύτρια και τους ομιλητές. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή και αν μπορούμε να εκπληρώσουμε τους στόχους της, πιστεύω ότι θα είμαστε και πολύ κοντά στην επιτυχία. Για διάφορους λόγους έχασε ανταγωνιστικότητα η Ευρώπη, χάσαμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Πρέπει να το κερδίσουμε ξανά και αυτό μπορεί να γίνει με απλές και λογικές προτάσεις και με επενδύσεις. Και θα ακολουθήσει ο ιδιωτικός τομέας, θα έχουμε λοιπόν επενδύσεις στην Ευρώπη. Συμφωνώ απόλυτα ότι χρειαζόμαστε ε, πράσινη ε, επανεκβιομηχάνηση καθώς και περισσότερες συνέργειες, ε, καλύτερη και περισσότερη υποστήριξη, ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, ε, τα τεχνικά, τεχνολογικά ιδρύματα. Υπάρχει περίπτωση ε, πολλά από αυτά να κλείσουν. Θα πρέπει να στηρίξουμε όμως τις μικρές ενωσιστηθήσεις επιχειρήσεις, τα εκολαπτήρια επιχειρήσεων και ήμουν πολύ ευτυχή γιατί γύθηκα μια επιτροπή ε, μια αντιπροσωπεία που πήγαμε στο Βερολίνο τη Δευτέρα και την Τρίτη. Και εκεί είδαμε πολύ πρακτικά παραδείγματα των σχέσεων μεταξύ των πανεπιστημίων και αυτών των λεγόμενων κολαπτηρίων. Ε, και μετά πήγαμε και είδαμε και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ακριβώς λόγω των συνεργειών που υπάρχουν και επειδή υπάρχουν λογικές, πρακτικές πολιτικές, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια 468 νέες εταιρείες που συστάθηκαν, 10 μόνο από αυτές απέτυχαν, οι περισσότερες ε, λειτουργούν. Πρέπει λοιπόν να δούμε πού ε, έχουμε επιτυχίες και εδώ και αλλού και κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξασφαλίσει προστέμενη αξία ε, και βέλτιστες πρακτικές που να μπορέσει να εφαρμόσει και αλλού. Πραγματικά στο Βερολίνο ήμουν πάρα πολύ τυχερός ε, που κατάφερα να δω αυτά τα πράγματα και μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να τα επαναλάβουμε και αλλού. Και αυτό άλλωστε είναι και το πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι στηρίζω λοιπόν την έκθεση, χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις εργασίας, χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Και νομίζω ότι μπορούμε και εμείς ε, με τις αρμοδιότητες που έχουμε να βάλουμε το λιθαράκι μας. Πρόεδρος, α, με συγχωρείτε, Μαρή Τερέ, Σάντσε Σμιτ και άλλοι. Ίσως όμως και Μανέσκου πρώτα που θα εκπροσωπήσει τον Νότσι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Όχι μόνο σήμερα ε, που ζούμε μια περίοδο κρίσης, αλλά και γενικότερα για το μέλλον ε, των ε, οικονομιών και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Βλέποντας τα μέτρα, τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν για την επίτευξη του στόχου 2020 για ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας, για ανταγωνιστικότητα. Νομίζω ότι οι κράτη-μέλη μπορούν πράγματι να προχωρήσουν σε αυτές τις πολύ καλές δράσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε παραπάνω προσπάθειες στο πεδίο αυτό. Ορισμένα μέσα που μπορούν να βοηθήσουν για την επανεκβιομηχάνηση θα μπορούσαν να είναι κάποια νέα μέσα για την ανταγωνιστικότητα, όπως το νέο χρηματοδοτικό μέσο ή τα νέα χρηματοδοτικά μέσα που θα μπορούσε να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Κομισιόν και τα διορθωτικά ταμεία. Υπάρχει έρευνα και ανάπτυξη που μπορεί να φέρει προστέμενη αξία η ευφύης εξειδίκευση. Πρέπει να στηριχθούν επίσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο Σον Κέλλη το ανέφερε. Επίσης, καλύτερη συμμετοχή του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου, γιατί χρειάζεται καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερη υποστήριξη των τοπικών επιχειρηματιών των ΜΜΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και βέβαια μέσω της εκπαίδευση, μέσω της επαγγελματική κατάρτισης, με τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ ερευνητικών κέντρων και ιδιωτικού τομέα. Έτσι θα υπάρξει αυτή η ευφύς εξειδίκευση. Και ένα τεράστιο δυναμικό που μπορεί να προσφέρει έρευνα στον ιδιωτικό τομέα, στην βιομηχανία. Έτσι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Η έκθεση αυτή λοιπόν είναι σημαντική και τώρα στο πλαίσιο του νέου πακέτου και της νέας περίοδου προγραμματισμού νομίζω ότι είναι σημαντικό να εστιάσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι με τον τρόπο αυτό θα έχουμε περισσότερη οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες και πιο βιώσιμες ε, θέσεις εργασίας. Έξω και στηρίζω ε, τις προτάσεις της Γήτριας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Μαρή Τερέ, Σμίτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη Μαρία για την γνωμοδότησή της. Έχει στοχεύσει σε συγκεκριμένους στόχους και εμείς πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Η Επιτροπή μας έχει ασχοληθεί με τα θέματα της εκβιομηχάνησης. Ψηφίσαμε τον προηγούμενο Μάιο στην Ολομέλεια, σας θυμίζω. Ο βιομηχανικός τομέας, ο οποίος υποχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την οικονομική κρίση η βιομηχανική παραγωγή έχει μειωθεί περνώντας από το 20% στο 16% του κοινοτικού ΑΕΠ από το 2008 μέχρι το 2011 και έχει μειωθεί η απασχόληση κατά 11% στον τομέα. Συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στις υπηρεσίες, αλλά 80% των καινοτομιών και 76% των εξαγωγών προέρχονται από, από τη βιομηχανία. Για 100 θέσεις που δημιουργούνται στη βιομηχανία δημιουργούνται άλλες 60 με 100 στην υπόλοιπη οικονομία. Για κάθε βιομηχανική θέση ε, απασχόλησης ιδρύονται δύο, δημιουργούνται δύο στον τομέα των υπηρεσιών. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από μια βιομηχανική πολιτική κοινοτική και από όχι από 27 εθνικές, σε στενή όμως συνεργασία με το τοπικό και περιφερικό επίπεδο. Υπάρχουν και οι προκλήσεις επίσης ε, του αναπροσανατολισμού των βιομηχανικών ε, πολιτικών που είναι ένα θέμα θα έλεγα διαμεθοριακό στον τομέα της καινοτομίας, της κατάρκεσης, της αποκατάστασης του περιβάλλοντος και ελκυστικότητας της υπαίθρου. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου γιατί το δυναμικό των δημιουργικών και φάνταστων βιομηχανικών δραστηριοτήτων δεν λαμβάνονται υπόψη ουσιαστικά. Η Επιτροπή Πολιτισμού ψήφισε την έκθεσή μου για τις δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. 4% του κοινοτικού ΑΕΠ και 7 εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης ανήκουν στον τομέα αυτό. Είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται γρήγορα και προοδεύει συνεχώς. Είναι πλεονέκτημα για την απασχόληση, ιδιαίτερα για την απασχόληση των νέων. Οι βιομηχανικές στρατηγικές θα πρέπει να συμβαδίζουν με μια προσαρμογή των συστημάτων κατάρτισης, με μια γυτνίαση ανάμεσα στην κατάρτιση και την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα στον τομέα της βιομηχανίας. Μποστινάρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι, έρχεται σε πάρα πολύ καλό χρονικό στιγμίο, σε πολύ καλή χρονική στιγμή. Η Επιτροπή μας είναι πολύ φυσικό να μην είναι σε θέση από μόνη της να συζητήσει τα θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε αν θέλετε το θέμα αυτό με μια ευρύτερη στρατηγική που αφορά την οικονομία την ευρωπαϊκή. Δεν μιλάμε για ε, οποιασδήποτε μορφής εκβιομηχάνηση, αλλά για μια εκβιομηχάνηση η οποία να είναι συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος πλέον. Όλοι οι αναλυτές ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης καταλήγουν στο ότι οι χώρες οι οποίες πηγαίνουν καλύτερα οικονομικά είναι αυτές οι οποίες έχουν υψηλή βιομηχανική απόδοση και δραστηριότητα. Έχουμε το παράδειγμα της Κίνας σε παγκόσμιο επίπεδο βέβαια η οποία έχει ενισχύσει το ρόλο της στην παγκόσμια σκηνή και στις διμερείς συναλλαγές, ενισχύοντας επίσης η Κίνα και την θέση της γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία. Και έχουμε και τη Γερμανία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια αντίστοιχη περίπτωση. Κατά τη διάρκεια της κρίσης η Γερμανία επηρεάστηκε πολύ λιγότερο από ό,τι άλλες χώρες από την κρίση χώρες οι οποίες είχαν και αυτές βιομηχανικό παρελθόν. Στα πλαίσια των ανταλλαγών ανάμεσα στις δύο αυτές χώρες βλέπουμε ορισμένες στατιστικές ε, τις οποίες μας δίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βλέπουμε ότι μία από τις επιπτώσεις της ε, ε, εκβιομηχάνηση είναι ότι η μόνη χώρα η οποία έχει θετικό ισοζύγιο στις εμπορικές της συναλλαγές με την Κίνα και όχι μόνο στο εμπόριο αλλά και στη βιομηχανία είναι η Γερμανία. Έχει, ένα, έχει 5 δις επιπλέον εξαγωγές προς την Κίνα. Άλλες χώρες έχουν πολύ ψηλότερα κέρδη βέβαια, πολύ ψηλότερα ελλείμματα όπως η Ολλανδία με 49 δις η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία είναι ακόμα πιο χαμηλά. Λοιπόν, τι μας δείχνουν όλες αυτές οι στατιστικές. Μας δείχνουν μια ε, βιομηχανική πολιτική η οποία επιτρέπει μερικές φορές την ενίσχυση της θέσης της Γερμανίας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόκειται για μια βέλτιστη πρακτική, γερμανική πρακτική και πρέπει να μάθουμε από αυτήν και να την εφαρμόσουμε και στον δικό μας τον τομέα οι συνάδελφοι οι οποίοι ε, διαπραγματεύονται το γενικό κανονισμό επιβάλλουν ε, μερικές φορές ορισμένες επιπτώσεις οικονομικές και πρόστιμα στις επιχειρήσεις οι οποίες αποφασίζουν να μετακινηθούν ε, ενώ έχουν βοηθηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, το θέμα είναι να δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ποια είναι η κατάσταση Βλέπουμε ότι στην Ανατολική Ευρώπη υπάρχει μια ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας, αλλά ταυτόχρονα σε κάποιες χώρες ε, υπάρχει αποβιομηχάνηση. Φεύγουν βιομηχανίες και πηγαίνουν όχι προς την Ανατολική Ευρώπη, αλλά προς την Κίνα, την Ινδία και αλλού. Η Ευρώπη λοιπόν σήμερα ε, έχει ένα έλλειμμα στον τομέα των βιομηχανικών πολιτικών η Ευρώπη έχει υποστεί μια τεράστια ήττα στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας. Έβλεπα προημερών τηλεόραση και είδα ένα νέο, μια έρευνα πάρα πολύ ιδιαίτερη θα έλεγα που αναφερόταν στα θέματα της φοροδιαφυγής και των απατών των οικονομικών στην Ευρώπη. Υπάρχουν στην Ήπειρό μας μαύρες τρύπες στον τομέα των φορολογικών παραδείσων, στον τομέα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Και αυτό οδηγεί σε ένα dumping ανάμεσα στις διάφορες χώρες οικονομικό. Υπάρχει ανταγωνισμός στο εσωτερικό λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Όχι μόνο δεν έχουμε μία λοιπόν ενιαία βιομηχανική πολιτική, αλλά έχουμε και ανταγωνισμό ανάμεσα στις χώρες, κάτι το οποίο οδηγεί σε απώλεια θέσεων ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια σκηνή. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε την έρευνα και την ανάπτυξη. Υπάρχει μια πρόταση από πλευράς του Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει σαν στόχο την ενίσχυση και την αύξηση των επενδύσεων στον τομέα αυτό, γιατί οι τάσεις που ακολουθούμε εμείς είναι αντίθετες από ό,τι σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εξακολουθούν να αυξάνουν τις επενδύσεις τους. Η Κίνα είχε πέρυσι 7 εκατομμύρια νέους ε, ε, πτυχιούχους πανεπιστημιακού επίπεδου οι οποίοι προσελήφθησαν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο αυτό θα λειτουργήσει σαν πολλαπλασιαστή στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Αυτό θα λειτουργήσει σε ένα θετικό περιβάλλον για την οικονομία γενικότερα. Και εδώ πρέπει να έρθουμε σε κάτι που είπαν και οι προηγούμενοι. Small is beautiful, υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά είναι οι μικρές επιχειρήσεις ωραίες μεν, όμορφες μεν, αλλά και πιο εύθραστες και ευαίσθητες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν μια σωστή εταιρική σχέση με το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Ναι μεν το μικρό είναι και όμορφο, αλλά Παρακολουθούμε και τη δημιουργία υπερβολικά μεγάλων μορφών κονσόρτια τα οποία είναι ε, εξαιρετικές, εξαιρετικού μεγέθους και εξαιρετικής αποδοτικότητας. Πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε εμείς τέτοια οικονομικά σύνολα από την Κίνα και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ένα επιπλέον θέμα είναι το περιεχόμενο των εμπορικών ε, συμφωνιών τις οποίες συνάπτουμε και στην οποία θέλουμε να προχωρήσουμε στο τέλος του καλοκαιριού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έχει ε, ενημερώσει σωστά για την συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε ή για τη συμφωνία ε, με, στον τομέα των επενδύσεων με την Κίνα και με άλλες συμφωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις χωρίς να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα λόγω των επερχόμενων ευρωεκλογών, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα επηρεαστεί αρνητικά. Δεν αναφέρομαι εδώ σε θέματα που έχουν σχέση ε, με τον προστατευτισμό. Η χώρα μου είναι αλήθεια, ε, είναι μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει τη μάστιγα της φτώχειας θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταγωνίζεται στο διεθνές επίπεδο όχι μόνο σε συγκεκριμένους τομείς περιορισμένου μεγέθους, αλλά σαν ένας συνολικά τεράστιος οικονομικός παίκτη. Το στρατηγικό όραμα το οποίο έχουμε μέχρι τώρα δεν μας βοηθά. Λυπάμαι αλλά μακρηγόρησα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Λαμπέρ δύο παρατηρήσεις, δύο-τρεις. Ε, σημείωσα σοξιοπερίεργο αυτό που είπε ο κύριος Μποστινάρου για τους Ολλανδούς. Δεν κατάλαβα. Ο κύριος Μποστινάρου εκτός μικροφώνου. Ο, α, οι επενδύσεις λέει ο κύριος Φανίστελ Ρόε. Είπατε, νόμιζα ότι είπατε, ότι το ισοζύγιο πληρωμών ήταν αρνητικό. Ότι ήμασταν μια χώρα που έχει όπου έχει σημειωθεί επιβράδυνση. Ίσως επειδή έχουμε το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Τι σημαίνει δηλαδή. Πολλά αγαθά αποβιβάζονται, εκφορτώνονται στο ε, λιμάνι. Εκεί ε, καταγράφεται η εκφόρτωσή τους και μετά ε, διανέμονται σε όλη την Ευρώπη. Ναι μεν εκφορτώνονται και καταγράφονται στην Ολλανδία αλλά μετά ε, μεταφέρονται στη Γερμανία, στη Γαλλία κτλ. Άρα μην εμπιστεύεστε έτσι τα στοιχεία όπως ε, τα ακούτε. Δεύτερον, έτσι εμφανίζουμε εμείς τεράστιες εισαγωγές. Το θέμα λοιπόν δεν είναι ότι καταργούνται οι βιομηχανίες μας, αλλά επίσης επιστρέφουν κάποιες υψηλής τεχνολογίας θέσεις εργασίας. Αυτό δεν σημαίνει πολλές θέσεις απασχόλησης αμέσως, αλλά ε, σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο υψηλό επίπεδο γνώσης και τεχνολογίας. Ε, για παράδειγμα έχουμε πολύ ρομποτική, έχουμε υψηλού επίπεδου ρομποτικά συστήματα για λεωφορεία και άλλα που γίνονται από ρομπότ. Έτσι επανέρχεται παραγωγή από άλλα τμήματα του κόσμου στην Ευρώπη. Τέτοιου τύπου στατιστικές πρέπει να κοιτάξουμε. Κάτι άλλο υπόθηκε και από τον κύριο Ματούλα. Να αναφερθούμε σε αυτές τις ε, τεχνολογίες κλειδιά γενικής εφαρμογής, όπου είμαστε ηγέτες στην έρευνα, αλλά ουραγοί στην εφαρμογή. Βεβαίως, καλό είναι να υπάρχει πλαίσιο έρευνας, αλλά ε, τα ωφέλη τα δρέπουν οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ιαπωνία. Και τώρα περνάμε στην ανοτεχνολογία, στην ε, ε, οικονομία που βασίζεται στην ε, βιολογία, στην βιοοικονομία. Εάν όλοι αυτοί οι τομείς πρέπει να κάνουμε προσπάθεια για να μείνουν στην Ευρώπη. Ή το χρησιμοποιείς ή το χάνεις. Use it or lose it. Άρα να αναφερθούμε και σε αυτά που είπε ο Ταγιάννη πρόσφατα για τη βιομηχανία αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα τέτοια σημεία. Τέλος, για το 5. Χαίρομαι που το, που το αναφέρατε. Χρειάζεται μια στρατηγική για περαιτέρω εξειδίκευση. Αλλά γενικά, στο εσωτερικό κάποιων χωρών Υπάρχουν ε, νέες ε, συγκεντρώσεις ε, πρωτοβουλειών που μπορεί να προκύψουν από τις συμφωνίες εταιρική σχέσης τα επόμενα χρόνια. Αλλά δεν βλέπω σχέσεις μεταξύ διαφορετικών περιφερειών, γιατί αυτό επιτρέπει από τους μεν να μάθουν από τους δε. Αυτές οι νέες δυνατότητες θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι να περιορίζονται σε κάποια χώρα, κάποια περιφέρεια. Έτσι θα έχουμε ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία πάνω από αυτήν που σημειώνεται σε περιφέρειες, χώρες, πόλεις μόνο. Πριν από δύο μήνες ήμουν στην Κίνα και ζήτησα όταν πήγα σε μια μεγάλη κρατικά επιδοτούμενη εταιρεία και μου είπαν η Ευρώπη είναι πολύ επίπεδη. Τι εννοούσαν, ότι δεν ε, συζητούν για συνολικά τι πρέπει να γίνει για όλη τη χώρα. Ο καθένας παίρνει το κομμάτι του της πίτας, αλλά δεν συζητάνε πώς θα μεγαλώσει συνολικά η πίτα. Άρα, επειδή δεν είναι δυνατόν κάθε χώρα να έχει όλες τις υψηλού επίπεδου πρωτοβουλίες για τη βιομηχάνηση, πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπαθίες μας. Για παράδειγμα, για την ε, νανοτεχνολογία, Υπάρχουν 4-5 μεγάλα κέντρα που μας έχουν απομείνει επειδή τα υπόλοιπα έχουν πάει στην Ασία. Αλλά 4-5 δεν είναι τόσο λίγα. Θα μπορούσαμε να κρατήσουμε την ε, ε, πρωτοπορία μας. Να πούμε λοιπόν στις χώρες, κάντε επιλογές, επενδύστε σε ορισμένους τομείς, αλλά τα ωφέλη να διαδίδονται σε άλλες χώρες, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε νέες επιχειρήσεις που ξεκινάνε. Όλα αυτά ίσως θα μπορούσαμε να τα συμπεριλάβουμε και θα εξετάσω το ενδεχόμενο υποβολή κάποιων τροπολογιών προ αυτήν την κατεύθυνση, αλλά είναι πολύ καλή βάση αυτή. Πρόεδρο, ε, ο τελευταίο ομιλητή ήταν αυτό. Δεν ξέρω αν Μαρία θέλει να μα πει κάτι ε, για να κλείσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Άκουσα όλες τις ε, προτάσει Οι περισσότερες είναι απόψει που τι συμμερίζομαι. Φυσικά δεν θα ασχοληθούμε με την ε, μεταφορά ε, επιχειρήσεων εκτός Ευρώπης. Αυτό πάει αλλού. Πρέπει να ασχοληθούμε με τις επιχειρήσεις, να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση, ε, να υπάρχει υπεύθυνη στάση, να ενισχύσουμε την καινοτομία, να ενισχύσουμε τους τομείς εχμής όπως οι νανοτεχνολογίες. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν και που δημιουργούν ανάπτυξη. Συμμερίζω την άποψη της Μαρίας Τερέσα για την ενίσχυση που πρέπει να δώσουμε στις δημιουργικές και πολιτιστικές επιχειρήσεις μας. Και ευχαριστώ για όλες τις απόψεις που ακούστηκαν και ελπίζω να βελτιώσουμε έτσι την έκθεση που είναι ε, δική μας ευθύνη να την κάνουμε, να την κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Με συγχωρείτε. Δεν είδα την... Ε, και τον Σάρφο Μάνκη που θέλει να μιλήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα με την ερμηνεία. Μουζουρ, Ζικά, Τέτσκο, Φουγκουέτο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 ότι πολλοί πανεπιστημιακοί, ξέρω εγώ, γνωρίζω πολλούς ε, πανεπιστημιακούς και ξέρω ότι δεν έχουν επαφή με τον κλάδο. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθεί σύνδεση και σχέσεις μεταξύ του πανεπιστημιακού και βιομηχανικού κόσμου. Εγώ ε, έχω τους συνεργάτες μου ε, που προσπαθούν να προωθήσουν αυτές τις σχέσεις μεταξύ πανεπιστημίων και του κλάδου. Και υπάρχουν κάποια προβλήματα στην ε, δημιουργία αυτών των σχέσεων. Διότι ξέρω ότι σε μια σειρά από χώρε, για παράδειγμα, οι μελέτε που ο κλάδο μπορεί να αναθέσει στα πανεπιστήμια δεν μπορούν να ε, μπουν στον ισολογισμό ω δαπάνε, στον ισολογισμό των επιχειρήσεων. Πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. Η μόνη απόφαση που πρέπει να πάρουμε, που δεν είναι και πολύ αισιόδοξη, είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Για λόγους που σχετίζονται με το χρονοδιάγραμμα για αυτήν την έκθεση, θα έχουμε μόνο μία μέρα για να υποβάλουμε τροπολογίες. Αύριο στις 12 λίγη η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Διότι πρέπει να ψηφίσουμε τον Ιούλιο. Σας παρακαλώ λοιπόν, κινητοποιηθείτε όσοι θέλετε να υποβάλλετε τροπολογίες. Ταχαίως. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στο τελευταίο θέμα στην ημέρησα διάταξη, που είναι η μελέτη που εκπώνησε η Γενική Διεύθυνση για την Περιφερειακή και Αστική Πολιτική, για την στέγαση, τις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ για την στέγαση. πώς προσπαθούν ε, σε ορισμένες ε, περιοχές στα προάστια των πόλεων οι παρεμβάσεις της ΕΤΠΑ ε, να βοηθήσουν τον, και την κοινωνική ενοποίηση. Θα μας μιλήσει πρώτα η Διευθύντρια, η κυρία Βίτσεβα. Ευχαριστώ πολύ. Με χαρά να σας παρουσιάσω σήμερα την εργασία της μελέτης αυτής, την οποία παρήγγειλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία του κυρίου Κουτσουλίνο. Είναι, εδώ έχουμε την τελική έκθεση για το πώς η παρεμβάσεις μας στον τομέα της στέγασης βοήθησαν την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την ε, βελτίωση της κατάστασης στις υποβαθμισμένες συνοικίες μέσω των παρεμβάσεων που κάναμε κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Η μελέτη λοιπόν αυτή έκανε πρώτα ε, αναθεώρηση της πολιτικής, μετά εξέτασε 10 προγράμματα σε διάφορα κράτη-μέλη. Στόχος μας ήταν στόχος μας, μας ήταν να έχουμε ε, τις αντιδράσεις και να συγκεντρωθούμε έτσι στις ε, καλύτερες πρακτικές και αφού συζητήσουμε ε, τα αποτελέσματα θα ενημερώσουμε τους εταίρους μας στις περιφέρειες ε, της πόλης για να γίνει η προπαρασκευή για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού για την ανάπλαση των αστικών περιοχών με τα λόγου γνώσεως. Να παρουσιάσω πρώτα απ' όλα την επιλεξιμότητα και πώς εξελίχθηκε η έννοια της εξελιξιμότητας στον τομέα αυτό κατά την περίοδο 7-13 για να ξέρετε σε ποιο νομικό πλαίσιο έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις. Και μετά θα δώσω το λόγο στους ε, εμπειρογνώμονές μας. Ήταν πολύ περιορισμένη η αρχική επιλεξιμότητα. Ο αρχικός κανονισμός είχε περιορίσει την επιλεξιμότητα μόνο στα νέα κράτη-μέλη που εντάχθηκαν μετά την 1η Πέμπτη του 2004 και μετά το πεδίο εφαρμογή ε, επεκτάθηκε δύο φορές, την 1η το 2009, όπου η γεωγραφική επιλεξιμότητα επεκτάθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη για προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας και τη χρήση ανανεωσίμων σε αστικές περιοχές. Και το 2010, επίσης για όλα τα κράτη-μέλη, ήδη ε, επεκτείναμε λοιπόν, μάλλον όχι ήδη, επεκτείναμε και στις περιθωριοποιημένες συνοικίες. Συμπεριλάβαμε λοιπόν και κριτήρια κοινωνικά απασχόλησης για κάποιες επενδύσεις στις υποδομές αυτές τις περιφερειοποιημένες περιοχές. Γιατί το κάναμε αυτό. Καταλάβαμε ότι μόνο οι παρεμβάσεις στον τομέα της στέγασης έχουν μόνιμο αντίκτυπο. Και μέσω του πιλωτικού προγράμματος το Κοινοβούλιο μας επέτρεψε να ε, συλλέξουμε τεκμηρίωση η οποία θα αξιοποιηθεί στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Κάτι ακόμη βάσει το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ανάκαμψης αλλάξαμε κάποιους κανόνες για τα όργανα χρηματοπιστωτικής ε, τεχνικής ε, λειτουργίας και θελήσαμε να συμπεριλάβουμε και τα προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας για τις ε, υπάρχουσες κατοικίες. Για τη νέα περίοδο προγραμματισμού συζητάμε ακόμη τι θα γίνει Έχουμε ήδη βέβαια κάποιους κανόνες για το πώς θα εντάξουμε τις στεγαστικές παρεμβάσεις στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Να δώσω τώρα το λόγο στον Τζον Ντότ και Γιάν Μάρτεν Ντεβέτ από το φορέα ΕΚΟΡΙΣ που θα μας παρουσιάσουν ε, τις ε, μελέτες πώς αντιμετωπίσαμε και εάν αντιμετωπίσαμε τις προκλήσεις και τι διδάγματα μπορούμε να εξαγάγουμε από την εργασία μας αυτή. Ευχαριστώ την Διευθύντρια. Έχουμε δύο εμπειρογνώμονες μαζί τους. για Μάρτεν ο πρώτος, εκορής διευθυντής και έχουμε επίσης ε, και τον Τζον Ντότο ο οποίος είναι υπεύθυνος έρευνας του εκορής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει πρώτο το λόγο. Γιάν Μάρτεν, Ντεβέτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τα κεντρικά ευρήματα μιας μελέτης που έγινε μαζί με τους φίλους του LSE και του Μητροπολιτικού Ινστιτούτου Έρευνας της Βουδαπέστης. Όταν ασχοληθήκαμε με ένα τέτοιο θέμα, το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο βέβαια, και έχοντας προετοιμάσει τη χθες το βράδυ την παρουσίαση, είδα το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος εδώ. Ευτυχώς ε, το άνοιξα και δεν ήταν πάρα πολύ ακριβό σε σχέση με το έσοδά μου. Θα πείτε ότι είμαι πλούσιος. Ε, δεν είμαι και πολύ πλούσιος γιατί πληρώνω πολλοί φόρους αλλά πληρώνω λίγο γιατί μένω σε ένα διαμέρισμα στις Βρυξέλλες με πάρα πολύ καλή μόνωση. Αυτό που βρήκαμε στην έρευνά μας λοιπόν είναι ότι όλο και περισσότεροι κάτοικοι της Ευρώπης έχουν προβλήματα στο να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους στον τομέα του ηλεκτρικού ρεύματος. Μιλάμε λοιπόν για φτώχεια στον τομέα της κατανάλωσης ρεύματος και ε, γενικότερα. Ξεκινήσαμε λοιπόν κατά την περίοδο 12-13. Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να ενημερώσουμε σωστά το τι συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο ε, και στις περιφέρειες όταν έχουν να επεξεργαστούν προγράμματα αναζωογόνησης, τα λέγαμε, κάποιων περιοχών κατοικίας. Προσπαθήσαμε να βρούμε ποιες είναι οι προκλήσεις για τέτοιου είδους προγράμματα και ποια είναι τα μαθήματα που μπορούμε να ε, βγάλουμε μέχρι τώρα. Υπήρξαν βασικά τρεις μεγάλες κεντρικές ερευνητικές ερωτήσεις με πλούσιο περιεχόμενο. Πρώτον, σε ποιο βαθμό υπάρχουν αποδείξεις ε, επενδύσεων στον τομέα αυτό που συνεισφέρουν στην αναζωογόνηση των αστικών περιοχών. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το ERDF και τα προγράμματα αντιμετωπίζουν τα θέματα της αηφορίας και πώς αυτοί οι δύο στόχοι, πρώτον της εξοικονόμησης ενέργειας από τη μία και κοινωνικών βελτιώσεων από την άλλη συνδέονται και σε ποιο βαθμό στην πρακτική συνδέονται. Το δεύτερο ερώτημα είναι ποιε είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην προπαρασκευή και εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων αναζωογόνησης των περιοχών. Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά στα πλαίσια της εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών και ποια είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της επιλογής τους. Και το τρίτο ερώτημα είναι σε τι μαθήματα, σε τι συμπεράσματα μπορούμε να καταλήξουμε από το ε, ισχύον ε, καθεστώς και ποιο θα είναι το πλαίσιο που θα βοηθήσει τέτοιου είδους προγράμματα στο μέλλον να είναι επιτυχή. Πώς προχωρήσαμε. Βασικά μελετήσαμε την υπάρχουσα γενικά τα υπάρχοντα στοιχεία και τις δημοσιεύσεις και μελετήσαμε σε βάθος 10 περιπτώσεις ε, ανάπλασης περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας είπατε να κοιτάξουμε πίσω από τους αριθμούς και αυτό κάναμε. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις τις οποίες θα αναφερθώ, ε, δαπανίσαμε μία εβδομάδα, δύο άτομα, πήραμε συνεντεύξεις, ε, ασχοληθήκαμε με ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων, επισκεφθήκαμε τα διαμερίσματα ε, και τις πολυκατοικίες στις οποίες κατοικούν. Μιλήσαμε με τους κατοίκους και όλους τους άλλους εμπλεκομένους. Δέκα λοιπόν μελέτες, ε, όλες μεταξύ τους διαφορετικές. Άμα δείτε στην πρώτη στήλη η γεωγραφική κάλυψη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο πήγαμε στο Merseyside και στο Χάλτον ε, στα πλαίσια του προγράμματος REACH το οποίο ε, προσπαθεί να ε, βελτιώσει τη ζήτηση από πλευράς των οικοκυριών για την εγκατάσταση μέτρων βελτίωσης της οικολογικής αποδοτικότητας των διαμερισμάτων. Συγκεκριμένη περίπτωση 2.000 διαμερίσματα. Μετά περάσαμε στη Γερμανία στην Γερμανία δεν είναι πάρα πολύ διαδεδομένες αυτές οι παρεμβάσεις, αλλά ακολουθεί μια ενιαία θα έλεγα αντιμετώπιση στην περίπτωση της πόλης του Κέμνιτς. Υπήρξε το θέμα της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών και της κοινωνικής θέρμανσης. Είπαμε επίσης, είδαμε στην Εσθονία, στο Ταλίν, την κοινωνική διάσταση, την ένταξη των κοινωνικών κατοικιών και των ορφανοτροφίων, και επίσης και την εισαγωγή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και την χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας. Το Καμπρέ στη Γαλλία, το Καρτιέ Λαφορέ όπου 446 διαμερίσματα κοινωνικής κατοικίας αντιμετώπισαν θέματα μείωσης της υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, βελτίωσης της ποιότητας της ζωής και ασφάλειας και την ίδια την εικόνα και τη φήμη της γειτονιάς του. στην Λετωνία το σύνολο της χώρας μας απασχόλησε, βελτίωση της αποδοτικότητας με τις πολυκατοικίες, στις πολυκατοικίες τις μεγάλες που υπάρχουν εκεί. Στην Ουγγαρία ασχοληθήκαμε με την περιφέρεια 21 της Βουδαπέστης. Στην περιοχή κοινωνικής κατοικίας του Άντι υπήρχαν πολλά προβλήματα. Ε, μιλάμε για μια κοινωνικά ευαίσθητη αναζωογόνηση ή ανάπλαση ε, και πήγαμε στο Μόστου στην Τσεχία, ε, στις περιφέρειες ε, Χάνοφ και Στόφσκι με την ανακαίνιση 10 μεγάλων πολυκατοικιών. Στο πεδεμόντιο της Ιταλίας υπήρξε ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας της κοινοτικής κατοικίας, ιδιαίτερα με κάποιες ειδικές κοινωνικές ομάδες όπως οι μονογονικές οικογένειες. Στην Λιθουανία το σύνολο της χώρας εξετάστηκε ε, και ε, μέσω της χρήσης ε, του Ταμείου Τζέσικα. Και τέλος το, στην Πολωνία, στο Σιέρατς, η κεντρική περιοχή της πόλης γύρω από την αγορά και την κεντρική πλατεία. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορετικά γεωγραφικά επίπεδα παρέμβασης σε κάθε περίπτωση. Όπως είπε και η διευθύντριά μας πριν από λίγο, το νομοθετικό πλαίσιο έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι αρχικά είχαμε συγκεντρώσει την προσοχή μας μόνο στα νέα κράτη-μέλη, το άρθρο 7,2, σε σχέση με τις υπάρχουσες κατοικίες και τα προγράμματα αφορούσαν και η επιλεξιμότητά τους αφορούσε μόνο ε, περιπτώσεις οικογενειών που ήταν ιδιοκτήτριες των ε, διαμερισμάτων τους. Ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με το θέμα της ενέργειας αλλά ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να δώσουμε και κίνητρα για τη δημιουργία τοπικής απασχόλησης. Από το 2010 έχουμε ε, να αντιμετωπίσουμε γενικότερα το θέμα της κατοικίας και των, περιφερει... των περιθωριοποιημένων οικογενειακών ομάδων. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, διαφορετικά όρια σε κάθε περίπτωση γεωγραφικά και χρονικά και σε σχέση με το, τις δυνατότητες που μπορεί να έχει το ERDF να χρησιμοποιηθεί. Το 2% σαν παράδειγμα ή το 3% σε επίπεδο μεμονωμένων προγραμμάτων 4% ε, προσετέθη ε, και θα μπορούσαμε προσθέτοντας τα ποσοστά αυτά να φτάσουμε το 2015 στο 6% ενώ για κάποιες χώρες παραμένουμε στο 4%. Λοιπόν, το θέμα είναι πόσα από τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν. Ε, δεν χρησιμοποιήθηκαν όλα. Οι τελευταίοι αριθμοί, αριθμοί τους οποίους έχουμε στην διάθεσή μας δείχνουν ότι μόνο το 1 με 2% του συνόλου του ERDF δόθηκε στα προγράμματα αυτά ανάπλασης των κεντρικών περιοχών των πόλεων. Γιατί, πρώτον γιατί υπήρξε πάρα πολύ λίγος χρόνος για να υπάρξει προσαρμογή στις αλλαγές της νομοθεσίας. Δεύτερον, απαιτείται πάρα πολύ χρόνος για τους κανονισμούς να φτάσουν στο επίπεδο, αν θέλετε, της τοπικής αυτοδιοίκησης και επίσης και στον τομέα της οικοδομής γενικότερα. Τα προγράμματα είχαν ήδη προχωρήσει όταν τέθηκε το θέμα της επιλεξιμότητας για μία επιπλέον φορά και κάποιες χώρες αποφάσισαν να μην δαπανίσουν ε, τα διαθέσιμα ποσά της πιστώσεις που είχαν στη διάθεσή τους για τις κοινωνικές κατοικίες. Για τις νέες χώρες και ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποιώ το επίθετο αυτό, η Ουγγαρία, Πολωνία, Ρωμανία και Σλοβακία είναι αυτές οι οποίες και σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστιαία έδωσαν πολύ μεγάλα ποσά. 100 με 200 εκατομμύρια για κάθε μία από τις χώρες αυτές. Για όλες τις υπόλοιπες, τις παλαιές, την Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο πρώτο μεγάλο θέμα το οποίο τίθεται Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντότ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τώρα το ενδιαφέρον ε, τμήμα. Τι μάθαμε. Αυτό που θέλουμε είναι η ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπλαση. Αυτό θέλαμε να βρούμε. Αυτό ήταν το Άγιο Δισκοπότερο που ψάχναμε. Το βρήκαμε. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο διότι λόγω των νομοθετικών διαδικασιών και του χρόνου εφαρμογή, τα προγράμματα ή μόλις τελείωναν που εξετάσαμε ή μόλις είχαν τελειώσει. Δεν ήμασταν λοιπόν σε θέση να δούμε μεγάλης διάστασης τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Κάναμε λοιπόν κάποιες ε, ε, προβλέψεις. Είδαμε πολύ ενδιαφέροντα όμως στοιχεία, πολύ ενδιαφέροντα διδάγματα για το μέλλον βγάλαμε. Ένα από τα βασικά διδάγματα που είναι κάτι που έχουμε πει και προηγούμενε χρονιές, είναι, είναι αν θέλετε να αντιμετωπίσετε αυτού που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, τις περιοχές, τους ανθρώπους, δεν χρειάζεστε μόνο ολοκληρωμένα, αλλά και πολύ στοχευμένα μέτρα. Είδαμε λοιπόν αυτές τις περιπτώσεις, είδαμε ότι κυρίως αφορούν ιδιωτικέ κατοικίε χωρί να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα συνολικά τη γειτονιά. Αυτά τα εθνικά προγράμματα δεν καταφέρνουν να πετύχουν τους πραγματικούς στόχους τις περιφέρειες. Ήταν ad hoc δηλαδή ποιος εποφελείτος στη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο όπου κυρίως ασχολούνται με τις κοινωνικές κατοικίες αλλά χωρίς πραγματικά ολοκληρωμένα προγράμματα. Ωραία. Ε, βοηθήσατε αυτούς που μένουν στις κοινωνικές κατοικίες άρα που έχουν ανάγκες. Αυτό δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει. Αλλά όπου υπήρχε νομοθεσία που ήθελε να αντιμετωπιστεί συνολικά μια γειτονιά, τότε όντως πραγματικά βελτιώνεται την κατάσταση αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, υποβαθμισμένες περιοχές, υποβαθμισμένε ε, συνθήκες ζωής. Αυτό μας απέδειξαν και οι προηγούμενες μελέτες που είχαν χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. Τι είδαμε λοιπόν ως ε, επιπτώσεις, ως αντίκτυπο. Ίσως να μην σας εκπλήσει ότι επειδή κυρίως ασχοληθήκαμε με τέτοια θέματα, αυτό που διαπιστώσαμε έχει να κάνει με την ενεργειακή απόδοση. Δεν σας μιλήσω τώρα για κιλοτόνους, κιλοβάτ και τέτοια, αλλά όπως βλέπετε, στην Εστονία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη ε, Λετωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εδώ είχαμε προγράμματα, κυρίως ε, για την ενέργεια. Όλες οι δημοσιεύσεις και η προηγούμενη έρευνα καταδεικνύουν ότι αυτό έχει βέβαια κοινωνικά και οικονομικά θετικά αποτελέσματα. Αλλά είμαστε τώρα ε, στη μέση της διαδικασίας για να δούμε πώς ακριβώς θα επηρεάσει το πραγματικό εισόδημα τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά ε, προβλέπουμε ότι αυτό θα συμβεί. Αντιμετώπιση της, ε, του κοινωνικού αποκλεισμού εάν ε, βάλουμε α, β ή γ θα ήταν β ο βαθμός που θα βάζαμε. Στην ε, Τσεχία είχαμε προγράμματα και ήπια και σκληρά και προγράμματα του κοινωνικού και του ΕΤΠΑ για ε, κοινωνικές κατοικίες στον Ρώμα. Εδώ όντως συνέβαλε το ΕΤΠΑ θετικά. Το ίδιο και στην Εστονία, όπου δεν ήταν θέμα ΕΤΠΑ, ε, συγγνώμη, όπου αν δεν ήταν ε, το ΕΤΠΑ δεν θα κατάφερναν ε, οι νηπιακοί και ευρεφικοί σταθμοί να είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε. Στη Γαλλία ίσως είναι λίγο πιο άειλο αφορά την εικόνα που δίνουν οι περιοχές. Έχει να κάνει όμως αυτό με βελτιώσεις στην ποιότητα της ζωής, στο βιωτικό επίπεδο. Στη Γερμανία, αν και δεν πήγαν άμεσα οι πόροι του ΕΤΠΑ για την στέγαση, ήταν στα πλαίσια ενός γενικότερου πιο ολοκληρωμένου προγράμματος. Είδαμε βελτίωση της, ε, του επίπεδου ζωής σε περιοχές που ήταν πολύ υποβαθμισμένες. Στην Ιταλία, μέσω της διαδικασίας εφαρμογής, είδαμε ότι οι ένικοι συνεργάστηκαν και εργάστηκαν με διάφορους φορείς. Δημιουργήθηκε μια αίσθηση κοινότητας. Αυτό θα μπορούσε να έχει τεράστια επίπτωση στο μέλλον αυτών των κοινοτήτων. Και τέλος, Πολωνία. Το αντίθετο. Όπως το διαβάζω λοιπόν, η ε, ανάπλαση κάποιων πλατιών δεν βοήθησε στην ε, αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού διότι ε, αφαιρέθηκαν οι κάτοικοι, έφυγαν οι κάτοικοι, μετακινήθηκαν. Εάν βελτιώνεις την κατάσταση μιας περιοχής αλλά αφαιρείς τους κατοίκους, μετακινείς τους κατοίκους, είναι αντιπαραγωγικό αν κάναμε μελέτη στην Αμερική υπάρχουν ε, πολλά ε, προγράμματα που είχαν το, τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι μόνο θέμα Πολωνίας. Οικονομικές επιπτώσεις δεν είναι τόσο ε, μεγάλες. Εγώ μελετώντας επιτόπου τις οικονομικές επιπτώσεις περίμενα να δω κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά καθόλου δημιουργία δεξιοτήτων και θέσεων απασχόλησης. Περιμένεις να δεις κάτι τέτοιο. Αλλά όταν χτίσει ένα σπίτι, δημιουργείς εργασίες Έτσι περιμένει. Έτσι λέει η έρευνα. Αλλά το βασικό θέμα είναι πώ θα μετρήσει τον αντίκτυπο, πώ θα βελτιώσει τον αντίκτυπο για την περιοχή, την πόλη, την περιφέρεια. Και διαπιστώσαμε ότι τα προγράμματα κατάρτισης ήταν τμήμα του συνολικού τμήματος στη Γαλλία, την Ιταλία σε άλλες χώρες ε, ήταν μια αυτόματη ε, διαδικασία της αγοράς. Υπήρχαν στην Τσεχία και στην Ουγγαρία συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματική κατάρτισης πολύ ενδιαφέροντα όπου αλλάζουμε τις υποδομές και έτσι βελτιώνουμε τις ανάγκες για υπηρεσίες είτε είναι για νοσοκόμες είτε για ανθρώπους που ε, λειτουργούν μικρά κοινωνικά κέντρα και αν μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα τα άτομα αυτά είναι θετικό η ενθάρρυνση της ανάπτυξης ε, στις τοπικές οικονομίες σε γειτονιές. Αυτό ήταν ακριβώς ε, ο βασικός μας στόχος, να έχουμε προγράμματα του κοινωνικού ταμείου που μαζί με άλλα περιβαλλοντικά να βοηθήσουν. Συμβαίνει. Στο Ενωμένο Βασίλειο θέλαμε να ε, δημιουργηθεί μια τοπική αλυσίδα παράδοσης Προσθέσαμε λοιπόν, εκτιμούμε 5 εκατομμύρια ή 6 εκατομμύρια. Ό,τι και αν προστίθεται θεωρούμε τις ε, εκτιμήσεις μας, το μετρήσαμε και ήταν θετικό. Στη Λιθουανία πάνω από 50% των ε, εργασιών μόνωσης έγινε από τοπικές εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε οικονομική επίπτωση για την ε, περιοχή παρέμβασης. Αλλά αν εξετάσουμε λοιπόν τις μελέτες αυτών των περιπτώσεων, των συγκεκριμένων προγραμμάτων, βλέπουμε ότι κυρίως ήταν στο κέντρο αυτές τις προσπάθειες στην Τσεχία, τη Γερμανία και τον Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιφατικά λοιπόν στοιχεία και μερικά θετικά αλλά και κάποια αρνητικά διότι υπήρξαν πολλά προβλήματα στη διαδικασία διότι τα προγράμματα δεν αντιμετωπίζονται με ολοκληρωμένη άποψη δεν βοηθάνε ευρύτερες ε, ε, κοινωνικές θετικές επιπτώσεις. Όπως είπα, είναι περιορισμένη η οικονομική επίπτωση. Αυτά τα προγράμματα είτε λόγου σχεδιασμού, λόγω χρόνου διάρκειας, λόγω ικανοτήτων, λόγω γνώσης δεν μεγιστοποιούν τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που θα μπορούσαμε να είχαμε μόνο και από το ότι έχουμε στα σπίτια μας καλύτερη μόνωση. Αν με αυτόν τον τρόπο αναπτυχθούν δεξιότητες, ε, υπάρξουν τοπικές θέσεις εργασίας, αυτό έχει ευρύτερη επίπτωση. Κάτι που είδαμε σχεδόν σε όλα τα προγράμματα. Δεν υπήρχε ε, δυνατότητα μέτρησης των ευρύτερων κοινωνικών ωφελών. Ε, είδαμε χιλιοτόνους, είδαμε κιλοβάτα, αλλά δεν είδαμε πόσες θέσεις εργασίας τοπικά. Τι ποσοστό επιπλέον εισοδήματος στην περιοχή. Πόσα άτομα ε, βρίσκουν καλύτερη κοινωνική κατοικία. Άρα αυτό λείπει. Πρέπει να το καλύψουμε για να βελτιώσουμε την απόδοση των προγραμμάτων στο μέλλον. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει ότι τα προγράμματα στέγασης γίνονται από το κατασκευαστικό κλάδο. Έτσι δεν είναι. Δεν θα θέλαμε ειδικού από τις μεταφορές να ασχολούνται με αυτά. Αλλά αν θέλουμε ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, οι επικεφαλείς των προγραμμάτων πρέπει να έχουν ευρύτερη κατανόηση και γνώση. Και συναντηθήκαμε με πολύ ικανούς, με πολύ καινοτόμους ε, ανθρώπους, που, εργολάβους, που όμως ασχολούνται με ε, τις κατασκευές. Και δεν ξέρουν πολλά για το τι είναι και πώς λειτουργεί το κοινωνικό ταμείο. Πώς θα βελτιωθεί η επίπτωση της κοινωνική συνοχή της στέγασης. Όλα αυτά είναι θεωρητικά για τους εργολάβους. Εδώ υπάρχει έλλειψη στην αγορά και επίσης και οριζόντια ε, ενοποίηση αναθεματικό τομέα. Αυτό επίσης ε, εμποδίζεται από την έλλειψη γενικότερης γνώσης. Υπάρχουν και άλλες αδυναμίες. Καλό πρόγραμμα για στέγαση, αλλά υπάρχουν και άλλες αδυναμίες. Οι περιοχές παρέμβασης. Ήταν συγκεκριμένες ε, πολυκατοικίες ή συγκεκριμένες ε, περιοχές με ορισμένες ε, ε, κοινωνικές κατοικίες εποφελούνται τα άτομα που μένουν εκεί. Ε, Βεβαίω βελτιώνονται τα διαμέρισματά του. Αν τι γίνεται στην πλανή πολυκατοικία, χρειάζεται περισσότερη επένδυση. Είναι θέμα προγραμματισμού. Αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα. Επίση δεν μα εκπλήσει ολοκλήρωση, ενοποιημένη αντίληψη διαπιστώνεται εκεί που ήδη υπήρχε γνώση και πείρα τέτοια αντιμετώπισης. Άρα πρέπει να αλλάξει η αντιμετώπιση, να γίνονται ευρύτερα γνωστές οι καλύτερες πρακτικές κτλ. Χρηματοδότηση βέβαια είναι αναγκαία για όλα. Και λόγω της συγκυρία ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει. Άρα δεν μας εκπλήσει και εδώ ότι επειδή το ποσοστό απορρόφησης του Τζέσικα, γιατί κυρίως τα ε, κονδύλια του ΕΤΠΑ κυρίως απορροφούνται, το Τζέσικα χρησιμοποιήθηκε όμως και αυτό από τις μελέτες που κάναμε είδαμε ότι αυτή η ιδέα τα δάνεια να δίνονται στους τελικούς χρήστες, σε άτομα συγκεκριμένα ή σε ομάδες τοπικές, τι θέτει το θέμα ποιος λαμβάνει τα χρήματα, πώς τα αξιοποιεί. Πολλές φορές χρειάζονται ε, ορισμένες οργανώσεις, αυτοργάνωση δηλαδή των κατοίκων. Αλλά αν κατέβει κανείς ε, πραγματικά στι πολυκατοικίε, τα άτομα που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη είναι τα άτομα που έχουν το μικρότερο επίπεδο, την μικρότερη δυνατότητα αυτοοργάνωση, την μικρότερη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν οι ίδιοι τα συμφέροντά του. Χρειάζονται στήριξη. Επίση χρειάζεται συγχρηματοδότηση ή δάνειοδότηση. Αλλά δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Εάν ε, θέλετε να δώσετε ένα δάνειο σε κάποιον για να βελτιώσει το, την μόνωσή του, υπάρχει ε, χαμηλή απορρόφηση γιατί δεν θέλουν να χρεωθούν, γιατί υπάρχει ανασφάλεια. Επίσης η χρηματοδότηση, δύσκολη. Οι τοπικές, οι περιφερειακές αρχές, άμα πάμε σε αυτές και τους πούμε ε, να δώσω το 50% μας λένε, μα τι μας λέτε τώρα, εμείς μόλις απολύσαμε χιλιά άτομα. Καινοτομία, ίσως δεν είναι η καλύτερη λέξη, αλλά χρειάζονται δυναμικοί τρόποι δυναμική τρόπη χρηματοδότηση. Η Τζέσικα ίσω είναι μια καλή αρχή, ίσω όμω χρειάζεται μια νέα αρχή την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Είναι σημαντική λοιπόν η συμμετοχή των χρηστών. Πρέπει οπωσδήποτε οι ένικοι, όσοι μένουν ευρύτερα στην περιοχή να συμμετάσχουν. Έχουν όμω σημειωθεί τεράστιε διαφορέ σε ορισμένε χώρε. Έχουμε κοινοτικά φόρουμ, ε, τοπικά φόρουμ, έχουμε ομάδε χρηματοδότηση όπω στη Γερμανία. Σε άλλε απλώ διαβούλευση. Ορίστε τα προγράμματα, ποια είναι η γνώμη σα Πέντε λεπτά, ορίστε, ευχαριστώ πολύ. Α αρχίσουμε να σκάβουμε. Καλύτερε πρακτικέ, να καταλάβουμε, να καταλάβουμε οι εργολάβοι, να καταλάβουν αυτοί που κάνουν, αυτοί που χτίζουν, να καταλάβουν ότι αν μα ακούσουν, αν συλλέξουν ευρύτερη πληροφόρηση, μπορούν να τα κάνουν καλύτερα τα σπίτια. Η συμμετοχή είναι ισχυρότερη στην φάση του προγραμματισμού, όταν γίνονται τα αρχικά σχέδια, λένε τη γνώμη του, αλλά μετά όταν περνάμε στην, στην κατασκευή γίνονται προσαρμογέ, μεγάλε αλλαγέ χωρίς ουσιώδη διαβούλευση του κοινού. Αυτό δημιουργεί δυσχέρες μετά, ώστε να δεχθεί τις αλλαγές, το κοινό, τις αλλαγές που γίνονται στο σπίτι τους μέσα, στο κατόφλι τους. Αλλά υπήρξε κάποια καινοτομία στο Ενωμένο Βασίλειο, υπήρξε η προσέγγιση ε, ανταγωνισμού, αλλά επίσης και καθορισμού ενός υπευθύνου ανά περιφέρεια, ο οποίος ε, εκλέγεται και μετά ε, ε, προωθεί τις αλλαγές. Αυτό ε, έκανε και άλλες περιοχές λίγο παρακάτω να θέλουν κάτι τέτοιο. Επίσης πρέπει να έχει λογικό κόστος η παρέμβαση. Το κόστος των ενεργειακών προσαρμογών στα σπίτια τονίστηκε. Ναι, έτσι κερδίζουν οι χρήστες διότι καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα. Αλλά αυτές τις εξοικονομήσεις τελικά τις παίρνουν οι χρήστες, οι ενοικιαστές, μπαίνουν στην τσέπη τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για πρώτη φορά για παράδειγμα μπήκαν ατομικοί μετρητές και αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκαν οι λογαριασμοί τους. Γιατί χρειάστηκε ε, να περάσουν μήνες μέχρι να καταλάβουν ότι τώρα που υπάρχουν ατομικοί μετρητές δεν πρέπει να αφήνουν συνέχεια αναμένα τα σώματα μέρα νύχτα. Άρα χρειάζεται ένα φυλάδιο να καταλάβουν δηλαδή τι σημαίνει ενεργειακή αποδοτικότητα, ποιότητα. Αντί να αξιοποιηθούν αυτές οι πιστώσεις του ΕΤΠΑ για να φτάσουμε στις καλύτερες, πιο σύγχρονες τεχνολογίες, υπήρξε μια πιο μετριοπαθής ε, προσέγγιση, γιατί θέλουμε να ε, βελτιώσουμε όσο περισσότερα κτίρια γίνεται. Αυτό είναι και θετικό, αλλά και πρόκληση. Το ΕΤΠΑ ποτέ δεν θα μπορέσει να πληρώσει για όλες τις τεραστικές παρεμβάσεις, Άρα πρέπει να πιέσουμε για περισσότερη καινοτομία. Αλλά εάν μπορούμε να ωφελήσουμε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, γιατί όχι. Ο τώρα, το λόγο στο Γιάννη για να σας ε, πει για τις ε, προκλήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εν να σα αναφέρω τι σημαντικότερε προκλήσει, Τι ανέφερε ο συναδελφό μου, αλλά μπορούμε να τι ομαδοποιήσουμε ενδεχομένω ω εξή. Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κρατικών φορέων, τοπικών αρχών, τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε γκάρσιο και σε οριζόντιο επίπεδο. Φυσικά αυτό το οποίο απαιτείται είναι περισσότεροι φορείς για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τέτοιες δράσεις, ιδίως εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε και μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και βέβαια σίγουρα απαιτείται στα διάφορα τομεακά σχέδια είτε αυτά είναι στον τομέα της στέγασης, είτε στον τομέα της ενέργειας, είτε της αποκατάστασης ή ανάπλαση σε όλα τα επίπεδα και σε εθνικό και σε τοπικό επαρχιακό θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση, πολύ σημαντική. Φαντάζομαι ότι έχετε συζητήσει σε εδώ και τη συμβατότητα των κανόνων και στόχων. Χρειάζεται λοιπόν και εδώ μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να γίνει και συσχετισμό του Κοινωνικού Ταμείου και του ΕΤΠΑ. Τέλο, πρέπει ε, να υπάρχει μια αναλογία τη χρηματοδότηση, μια αντιστοίχηση τη χρηματοδότηση ε, ανάλογα με τι ανάγκε λόγω και τη κρίση του κλίματο. Ε, θα πρέπει δηλαδή να εξετάσουμε τη δυνατότητα ε, το, της δανειοδότησης ε, ακόμη περισσότερο, παρότι και αν είναι περιορισμένες πλέον οι δυνατότητες ε, δανειοδοσίας. Έχουμε εστιάσει πολύ περισσότερο στο δημόσιο τομέα. Όμως ο ιδιωτικός τομέας καταλαμβάνει πολύ μεγάλο μερίδιο σε πολλά κράτη-μέλη. Και πιστεύω ότι εκεί έχουμε, μάλλον αυτό πρέπει να προσέξουμε ότι εκεί υπάρχουν κάποιες ενώσει οι ενώσει των ιδιοκτητών που πιο δύσκολα μπορεί κανείς ε, να τις διαχειριστεί για να πάρουν ε, στήριξη. Ε, υπάρχουν διάφορες διαδικασίες, είναι πιο δύσκολο, ιδίως βράχει πρόθεσμα. Η ηγεσία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική, η τοπική ηγεσία, είτε από κάποια ένωση ιδιοκτητών, είτε από κάποιο δήμο, αυτό πάντοτε ήταν σημαντικό. Σημειώσαμε επίσης τις προτάσεις ε, της Κομισιόν για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Οι προκλήσεις που βλέπουμε εδώ βλέπουμε ότι ε, αντιμετωπίζονται με τις προτάσεις της Κομισιόν. Έχουμε τις ταγαστικές παρεμβάσεις, οι οποίες εντάσσονται πολύ καλώς θεματικούς στόχους ε, που ε, συμπεριλήφθησαν και στη Συμφωνία Εστερικής Σχέσης. Τουλάχιστον τέσσερις από τους 11 θεματικούς στόχους καλύπτονται. Έχουν έμεση ή άμεση σχέση με τη στέγαση. Επίσης, δεν προτάθηκε κάποιο όριο ε, αφαιρέθηκε το όριο και αυτό είναι πολύ καλό για να μπορέσουν να γίνουν πιο ουσιαστικές επενδύσεις στον τομέα της στέγασης, στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ. Και επίσης ε, κάτι πολύ σημαντικό επιτόπου είναι να υπάρξει και μεγαλύτερη ευελιξία για τους ε, τύπους, τα είδη στεγαστικών δραστηριοτήτων. Ουσιαστικά υπάρχει ελευθερία. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αρκετές μορφές επενδύσεων. Σίγουρα καλό είναι και είναι δυνατόν να εστιάσει κανείς στην ενεργειακή απόδοση, στην κοινωνική συνιστόσα, όμως θα είναι ε, πιο ε, εύκολη και ισορροπημένη ε, προσέγγιση με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Θα συμπεριλάβουν και την πτυχή της καλύτερης δυνατότητας σύνδεσης. Βλέπετε, εν αυτό το τρίγωνο με τις τρεις διαστάσεις, ε, την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική. Και βλέπετε τις διάφορες θέσεις, τα τετραγωνίδια αυτά που δείχνουν ε, που πετύχαμε με τις παρεμβάσεις μας. Πρέπει να πει κανείς όμως ότι η χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων στέγασης μέσω του ΕΤΠΑ ε, κάνει τη διαφορά και πραγματικά έχει απτό αντίκτυπο σε μια σειρά από μέτωπα. Σίγουρα ισχυρότερος αντίκτυπος ήταν ε, στην ενεργειακή απόδοση, στην κοινωνική ένταξη, λιγότερο στην οικονομία. Γνωρίζουμε όμως ότι ε, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και για την ολοκληρωμένη προσέγγιση φυσικά χρειάζεται και ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο πολιτικής και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Πολύ σημαντικό το πόρισμα αυτό. Επίσης, η νέα περίοδος προγραμματισμού θα πρέπει να δώσει κίνητρα προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. προσέγγιση. Είμαστε ε, ε, μετριοπαθώς αισιόδοξοι, αλλά θεωρούμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, και το ζήτημα της φτώχειας και πιστεύω ότι με τι επενδύσει ε, του ΕΤΠΑ μπορούν να γίνουν πράγματα, αλλά σίγουρα το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί μόνο με αυτό. Uh, uh, Πρόεδρο, ευχαριστώ. Ποιοι να θέλουν να λάβουν το λόγο, η Μαρή Τερέ πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές, ήταν πληρέστατη παρουσίασή του και μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να συζητήσουμε πάρα πολύ ε, συγκεκριμένο αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και για το μέλλον της πολιτικής συνοχής που τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάρει μια εντονιαστική διάσταση ε, με την πρόθεση του Επιτρόπου βέβαια και χαίρομαι που βλέπω ότι και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού επίσης θα είναι μεγάλη αιστεία στον τομέα αυτό. Ξέρετε ότι ο πρώτος στόχος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνοχής είναι η ισορροπία ε, μεταξύ των εδαφών. Ξέρουμε ότι το 68% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε μετροπολιτικά κέντρα που αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το 70 περίπου του ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, 75% τη ενεργειακή κατανάλωση. και επομένω καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Και πρέπει να παρακολουθήσουμε και την εξέλιξη της αστική πολιτικής για να έχουμε το πρασίνισμα ε, των ευρωπαϊκών εδαφών. Θα ήθελα να κάνω κάποια ε, ερωτήματα. Ε, είπαμε 20 δις θα πρέπει να δοθούν για την αστική ανάπτυξη, μεγάλο δηλαδή κομμάτι του συνολικού προεπλισμού συνοχής. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάποια ιδέα για το ποσό αυτό, αν δηλαδή πανήθηκε ε, σωστά, αν πανήθηκαν αυτά τα ποσά, τι όγκους έχετε να μας αναφέρετε. Ποια ταμεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες συγκεκριμένα σήμερα ήδη μπορούμε να ξέρουμε την αναλογία, ε, τι κονδύλια θα πάνε προς την ε, αστική ανάπτυξη συγκεκριμένα. Και επίσης ένα άλλο σημείο που είναι ιδιαίτερα προσφυλές, επειδή είμαι από το Περπινιά, την Νότια Γαλλία, εκεί έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ιστορικό κέντρο, η παλιά πόλη, και η ανάπλαση ε, αυτού του ιστορικού κέντρου αποτελεί μείζωνα πρόκληση για το μέλλον. Το κέντρο της πόλης απειλείται όμως ε, επειδή δεν έχουν επενδυθεί αρκετοί πόροι. Επίσης ε, κλείνουν τα μαγαζιά στην περιοχή επειδή ε, δέχονται τον ανταγωνισμό της περιφέρειας, η ανακαίνιση είναι πολύ δύσκολη λόγω κάποιων αρχιτεκτονικών περιορισμών, υπάρχουν αθυγινές κατοικίες ή μη προσαρμοσμένες τουλάχιστον από ενεργειακής πλευράς, είναι πολλά αυτά τα κτίρια και άρα είναι ακατοίκητα, δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης, επαρκής τα μέσα συγκοινωνίας δεν έχουν φτάσει το μέγιστο ε, επίπεδο απόδοσης για να είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν στήριξη από το Ταμείο Συνοχής και με τα κονδύλια του ΕΤΠΑ Νέας Γενιάς ελπίζω να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες, να έχουμε την ολοκληρωμένη αυτή ανάπτυξη. Το 5% ε, του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ θα πάει σε αυτή την ε, συνιστόσα Ολοκληρωμένα λοιπόν συνολικά φαίνεται ότι το κέντρο, το ιστορικό κέντρο των πόλεων ε, φαίνεται να ωφελείται και σίγουρα θα πρέπει και οι τοπικοί αυτοδιοίκηση δήμοι ε, να επωφεληθούν και να ζητήσουν να ε, μπορέσουν να πάρουν στήριξη στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που βέβαια ακόμα υποσυζήτηση. συζήτηση. Εμείς οι, Ευρωπαίοι, οι Ευρωβουλευτές ξέρετε ότι πολλές φορές έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την έλλειψη προβολής ορατότητας ε, της προσθέμενης αξίας τέτοιων προγραμμάτων. Ε, πρέπει λοιπόν ε, και εσείς να κάνετε τη δική σας δουλειά και εμείς ως Ευρωβουλευτές έχουμε το δικό μας ρόλο. Σας ευχαριστώ για μια κομφέτα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη σας. Ο Γιάνν Όλμπριχτ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η έρευνα δείχνει ποιες είναι οι αδυναμίες στο σύστημα και οι πραγματικές προκλήσεις. Θυμάμαι ότι πριν το 2007 είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με το αν η κοινωνική κατοικία είναι ευρωπαϊκό θέμα ή όχι. Έγινε μια πολιτική συζήτηση και καταλήξαμε στο ότι δεν είναι. Και δεν θα πρέπει να υποστηρίζουμε την κατοικία γενικότερα γιατί σύμφωνα με την επικουρικότητα αυτό είναι θέμα δήμων, κοινοτήτων και η άλλη απάντηση είναι ότι αν πράγματι τα λάβουμε υπόψη μας αυτό αφορά τις δυνατότητες επένδυσης σε εθνικό επίπεδο, δημόσιες επενδύσεις, ιδιωτικές επενδύσεις, επιδοτήσεις από πλευράς των κρατικών υπηρεσιών Καμία σχέση όμως με τη Γενική Διεύθυνση ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, περισσότερο θέματα ανταγωνισμού είχαν τεθεί όταν ε, είχαν αναλυθεί κάποια παραδείγματα για την ανάπλαση κοινωνικής κατοικίας στην Ολλανδία και όλες αυτές οι συζητήσεις έδειξαν ότι δεν έχουμε μόνο να κάνουμε με με οικονομικά θέματα, αλλά έχουμε να κάνουμε με θέματα λίγο πιο περίπλοκα. Σαν παράδειγμα η κοινωνική κατοικία στις περισσότερες χώρες ελέγχεται και αναπτύσσεται, πολλές φορές γίνεται και αντικείμενο διαχείρισης από ιδιωτικές εταιρείες. Για ένα λοιπόν τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κοινωνική κατοικία είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Είναι θέμα καταπολέμησης ένδυας κτλ. Για ένα άλλο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κατοικία είναι θέμα ενεργειακής αποδοτικότητας. Εδώ συνδέονται και οι ερωτήσεις της Μαρή Τερέζ ε, σε σχέση με το πόσα χρήματα δαπανήθησαν. Είναι πάρα πολύ αργά γιατί να μάθουμε ακριβώς γιατί δεν είχαν καμία διάθεση να αναπρογραμματίσουν οι κρατικές υπηρεσίες στα συστήματά τους και τα συστήματα στα πλαίσια της κοινωνικής κατοικίας είναι πάρα πολύ ε, περίπλοκα. Κάποιοι χρησιμοποιούν και τα κριτήρια της ενεργειακής αποδοτικότητας. Άλλοι θεωρούν ότι το, πνεύμα το πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα του τομέα, της δραστηριότητας, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των οικοδομικών. Γιατί για πολλές χώρες και για άλλες οικονομίες βέβαια η κατοικία θεωρείται και η οικοδομή η κινητήρια δύναμη της οικονομίας τους, κάτι το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο σήμερα πια βέβαια, για το ποια είναι τα αποτελέσματα. Αυτή ήταν η συζήτηση που γινόταν το 2007. Η συζήτηση συνεχίζει να γίνεται. Πράγματι τα έχουμε ε, στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αυτά, αλλά κατά τομής όμως. Και ένα κομμάτι είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν θα πρέπει όμως να κρύβουμε ότι αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζει το σύνολο των παρεμβάσεών μας και στον τομέα των ταμείων συνοχής, του Ταμείου Συνοχής. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά εφόσον ε, ε, υπάρχει πολιτική συμφωνία, η κοινωνική κατοικία είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Εφόσον είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, Έχουμε ένα καλό παράδειγμα έτσι ώστε να δείξουμε ότι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση δεν είναι κάτι το θεωρητικό αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει με σωστό τρόπο διαφορετικές πολλαπλές μορφές χρηματοδότησης για πολλαπλούς στόχους οικονομικούς, κοινωνικούς κτλ. Πρέπει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παράδειγμα με σωστό τρόπο. Η έρευνά σας το δείχνει. Αλλά δεν θα πρέπει να μείνουμε σε επίπεδο αναγγελίας μόνο. Ίσως οι νέες μέθοδοι ε, για τα διαφορετικά ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το στοιχείο αυτό είναι πολυδιάστατο. Αλλιώς θα μείνουμε σε επίπεδο, ε, θα έλεγα, πολιτικών διακηρύξεων θα πρέπει να αναφερθούμε όχι μόνο σε κοινωνική κατοικία αλλά και στις ε, ιδιωτικές κατοικίες. Αν αυτό όμως το βάλουμε τότε θα έχουμε προβλήματα με τις επιδοτήσεις τις κρατικές. Μιλάμε για την ενεργειακή αποδοτικότητα, μιλάμε για τα κτίρια. Τα κτίρια δεν είναι μόνο η κατοικία, είναι κάτι και το εσωτερικό, είναι λίγο περίπλοκη η κατάσταση και κάθε κομμάτι αυτής της συζήτησης κρύβει και κάτι άλλο από πίσω. Δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε όλα αυτά πάρα πολύ εύκολα. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε μια αυτονομία ανάμεσα σε όλα αυτά. Είναι μια από τις λίγες δυνατότητες πάντως που έχουμε εδώ να χρησιμοποιήσουμε το σύνθημα που θέλουμε να χρησιμοποιούμε το της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Ιωακίμ. Ευχαριστώ και εγώ για την παρουσίασή σας, διότι αντιμετώπισε με κριτικό πνεύμα το θέμα και έκανε μία μελέτη που ε, διαφοροποιημένα εκτίμησε τα αποτελέσματα σε κάθε χώρα. <clears throat> Οπότε προέκυψε ότι δεν είναι μόνο θέμα βέβαια χρηματοδότησης, αλλά είναι και θέμα τρόπου εφαρμογής, στρατηγικής και συνεργασίας μεταξύ διαφόρων εμπλεκομένων. Και αυτό που είπε και η Μαρή Τερέζ, τα προβλήματα με την ανάπτυξη των πόλεων είναι πρόβλημα περιφερειακού επίπεδου. Εκεί γίνονται τα λάθη. Εκεί λαμβάνονται λάθος αποφάσεις. Και το ξέρω και από πολλέ ε, πόλεις στη Γερμανία, ιδίω στην Ανατολική Γερμανία. Αμέσως μετά την πολιτική αλλαγή δημιουργήθηκαν αυτά τα τεράστια εμπορικά κέντρα σε χώρους πρασίνου. Και οι υποβαθμισμένε συνοικίε δεν πήραν φράγκο από πλευρά δημιουργία επιχειρήσεων και υποδομών. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, από τη μία σε κάποιες περιοχές έχουμε ε, θαυμάσια ανακαινισμένα ιστορικά κέντρα, αλλά δεν υπάρχουν επιχειρήσεις εκεί και μαγαζιά. Γιατί έχουν γίνει αλλού τα μαγαζιά και είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτή μετά η αλλαγή γιατί λήφθηκε αρχικά μια πρώτη λανθασμένη απόφαση. ότι η στέγαση μετά την ε, διατροφή και την ένδυση είναι πολύ σημαντικός τομέας, είναι προφανές. Αλλά έχει δίκιο ο Γιάννα, αυτά ξεκινάνε συνήθως μέσω ιδιωτικών φορέων. Βεβαίως. Ακόμη και οι επιχειρήσεις για την ε, δημιουργία, για την κατασκευή κατοικιών σε επίπεδο ενός ε, Δήμου μπορεί να είναι ιδιωτική επιχείρηση και μετά πουλάνε ή νοικιάζουν αυτά τα διαμερίσματα και η συντήρηση της ε, ε, πολυκατοικίας είναι θέμα των ενοικιαστών, των κατοίκων, των ιδιοκτητών και αν θα τα πληρώσουν αυτά ή αν θα πρέπει να παρέμβουν ε, και οι δημόσιοι φορείς είναι θέμα συζητήσιμο, αλλά αρχικά είναι ιδιωτικό θέμα στη Γερμανία. Τα διαθροτικά ταμεία δεν συμβάλλουν στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, αλλά φυσικά έχουμε το πρόβλημα ότι κυρίως στις μεγάλες πόλεις, ε, αλλά ακόμη και στις μεσαίες πόλεις τώρα. Έχουμε ολόκληρες γειτονιές, όπου ε, υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα και αυτό αντανακλάται και στην ε, συνύπαρξη των ανθρώπων. Δεν μ' αρέσει που ε, αντιτίθεμαι σε αυτό που είπε η Μαρή Τερέζ. Οι πρώτοι που τόνισαν τα θέματα αυτά ήμασταν εμεί ω κοινοβούλιο Γιάνν Ολμπριχτ με το Intergroup για τα θέματα αυτά των πόλεων. Εμεί τα τονίσαμε. Τα συζητήσαμε ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από ό,τι θυμάμαι εγώ και από ό,τι μου είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, έτσι γινόταν πάντα. Τι χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα, να είναι διατεθειμένοι οι διάφοροι εμπλεκόμενοι, το είπατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα από κοινού, να συνεργαστούν. Και εμείς το μάθαμε αυτό στο Βερολίνο για, τα, για τις προβληματικές γειτονιές όπου υπάρχουν πολλοί μετανάστες, ε, διάφορες κοινότητες που δεν συνεργάζονται, υψηλή ανεργία, δύσκολες κοινωνικές σχέσεις. Εκεί επιλέξαμε την οδό τη διαχείριση σε επίπεδο γειτονιάς για να δημιουργηθεί, δημιουργηθεί μια κοινότητα, μια κοινή αντιμετώπιση. Αν βελτιώσουμε, διαπιστώσαμε τη στέγαση, τότε βελτιώνεται και η ατμόσφαιρα στη γειτονιά. Έτσι νομίζαμε. Αλλά μετά διαπιστώσαμε ότι δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει εάν δεν συμμετάσχουν οι κάτοικοι γιατί ε, το θεωρούν ότι είναι κάτι που τους επιβάλλεται απ' έξω με το οποίο δεν έχουν καμία σχέση αντίθετα φοβούνται ότι αν ε, ανακαινιστούν ε, οι κατοικίες θα τους διώξουν από τις γειτονιές αυτές θα έρθουν υψηλότερα αμοιβόμενοι να ζήσουν σε αυτές τις περιοχές πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες των διαφορετικών ταμείων με το κοινωνικό ταμείο όλοι αυτοί να συνεργαστούν με τους ε, κατοίκους ε, στις γειτονιές αυτές. Μόνο αυτό θα οδηγήσει σε επιτυχία. Ε, πριν από λίγες μέρες ήμασταν μια αντιπροσωπεία στο Βερολίνο και τους δείξαμε και μια τέτοια γειτονιά και πώς βελτιώθηκε. Αλλά οι διαδικασίες αυτές κρατάνε πάρα πολύ χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια αναβάθμιση μέσα σε τρία χρόνια. Αλλά δυστυχώς ε, οι διαδικασίες μας ε, προωθούν πιο πρόθεσμα προγράμματα από ό,τι μπορούμε εμείς να διαπιστώσουμε. Χρειαζόμαστε 7 με 10 χρόνια για μια περιοχή που είχε υποβαθμιστεί και άρα απομονωθεί να αναβαθμιστεί, να αναπλαστεί. Να ληφθεί λοιπόν και αυτό υπόψη, η διάσταση χρονική. Και αν μπορέσουμε να πείσουμε όλους που συμμετέχουν τις επιχειρήσεις εκεί, τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές, εάν όλοι αυτοί καταλάβουν και επιτύχουμε να συνεργαστούν, τότε σημειώνονται επιτυχίες. Και αυτό σημαίνει ότι εισραίει και νέος πληθυσμός. Ε, για παράδειγμα, φοιτητέ, καλλιτέχνες. Εάν, για παράδειγμα, σε μια περιοχή είχαμε πάρα πολλά, έως και 80% άδεια σπίτια, γιατί κανείς δεν ήθελε να πάει, καταφέραμε να πείσουμε του ε, ιδιοκτητέ να τα νοικιάσουν σε καλλιτέχνε, για παράδειγμα γιατί έχει αναβαθμιστεί η περιοχή. Όλα αυτά πρέπει να αποφασίζονται όμω επί τόπου. Και ωραία η ενεργητική αποτελεσματικότητα αλλά ξέρετε πόσο ανεβαίνουν εκθετικά οι τιμές ε, ε, των καυσίμων, τη ενέργεια. Άρα όσε εξοικονομήσει δεν φαίνονται γιατί τι τρώει η άνοδος των τιμών τη ενέργεια. Διαπιστώνουν στο τέλο λοιπόν δεν πληρώνουν λιγότερα, πληρώνουν και περισσότερα όπω αναφέρθηκε. Πρέπει λοιπόν να τους πείσουμε. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί όμως πολύ συχνά η ενεργειακή βελτίωση. Γιατί πολλές φορές είναι τόσο ετοιμόρροπα τα κτίρια που πρέπει πρώτα απ' όλα πριν να ασχοληθούμε με ενεργειακή απόδοση να ε, ανακαινήσουμε τα κτίρια. Όλα τα θέματα αυτά χαίρομαι που τα αναφέρατε. Τι μπορεί να κάνει περισσότερο η Ευρώπη να ευνοήσει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ χωρών, μεταξύ δήμων, ούτως ώστε οι θετικές εμπειρίες που έχουν γίνει σε μία περιοχή να μην χρειαστεί να ξαναγίνουν, να αξιοποιηθούν. Ο καθένας να εργάζεται με βάση τις ήδη αποδεδειγμένα σωστές πρακτικές. Μία ερώτηση. Πριν από δύο-τρία χρόνια είχαμε αποφασίσει να υπάρξει απευθείας στήριξη των πόλεων που έχουν ιδιαίτερα περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμού. Ρώμα ή στην περίπτωση της Βουλγαρίας η τουρκική μειονότητα. Εδώ και δύο-τρία χρόνια διαπιστώνουμε ότι έχουν γίνει ε, σημαντικές μεταναστευτικές ροές εντός της Ευρώπης. Και με βάση το Βερολίνο όπου μένω, πέρσι ήρθαν 40.000 Ρώμα και άλλες ομάδες πληθυσμού από την ε, χώρα προέλευσης τους υποθέτουμε ότι δεν θα επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους οι ε, άνθρωποι αυτοί. Αλλά αυτό μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα ένταξής τους. Γιατί ήδη είχαμε προβλήματα στις ε, γειτονιές όπου έμεναν όπου πηγαίνουν και τις είχαμε κάπως ε, αναβαθμίσει αυτές τις περιοχές αλλά τώρα χρειάζεται να γίνει περαιτέρω προσπάθεια. Και πρέπει οπωσδήποτε να ε, αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά εάν οι πόλεις από όπου προήλθαν ε, τα άτομα αυτά να τους βοηθήσουν να μείνουν εκεί παρά τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις Εφόσον λοιπόν δεν το επέτυχαν οι χώρες τους ε, αυτό, να δημιουργήσουν ε, βέβαια όχι μόνο ε, κατοικίες αλλά και θέσεις απασχόλησης, είναι ευρύτερο το πρόβλημα. Τότε πού θα βρούμε εμείς τα λεφτά για να κάνουμε εμείς αυτό που δεν έκανε κάνει εκείνοι. Θα πρέπει να γίνει μια κάποια ανακατονομή των πόρων. Για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε ένα τέτοιον διαστάσεων καθήκον. Κοιτάξτε, ήμουν πολύ επίοικη απέναντί σα, Γιώαχημ, αλλά δεν θα είμαι επίκη με του επόμενου. Πρέπει να φύγουμε σε 10 λεπτά και έχουν ζητήσει ακόμη τρία άτομα το λόγο και θέλουμε να ακούσουμε και τι απαντήσει και την κυρία Διευθύντρια. Παρακαλά, δύο λεπτά. Βίκτορ, Ραμόν και Νίκο. Δύο λεπτά ο καθένα. Μποστινάρο. Δεν με ικανοποιούν μόνο δύο λεπτά. Καλά δυόμιση λέει ο πρόεδρο. Καλά δυόμιση. Όταν ξεκίνησα να συντάσω την έκθεση για το Ταμείο Συνοχής είχα μόνο εμπειρικού τύπου θα έλεγα αγνώσεις σε σχέση με το Ταμείο. Αλλά βλέποντας το αποτέλεσμα της έρευνας και θέλω να συγχαρώ εδώ τους δύο ερευνητές με ικανοποιεί ιδιαίτερα. We succeeded something which was fully confirmed by the study. First, the need Αλλά γιατί πετύχαμε καταρχάς να δείξουμε ότι είναι σημαντική η ανάγκη για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής, σε συνδυασμό με το Ταμείο Συνοχής και το δικό μας Ταμείο, σε τομείς όπως η ενέργεια. Λοιπόν, αυτή η πολυμερής αντιμετώπιση είναι κάτι το δεδομένο. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε όχι μόνο το Περιφερειακό και το Ταμείο Συνοχής, αλλά και το Θεογκά και άλλα ταμεία, στα οποία ε, υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού τους τοπικά. Τέταρτον, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Από τη μία έχουμε τη δυνατότητα αυτή στα πλαίσια της περιφερειακής διαχείρισης του δικού μας ταμείου, αλλά φυσικά αυτό το περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται από τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Αυτό όμως επιτρέπει την άσκηση της λεγόμενης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Και τέλος, από τον Ιάν, χωρίς να είμαστε ιδιαίτερα οραματιστές, πετύχαμε να συνδυάσουμε κάποια σημαντικά πράγματα, όπως στην παραγωγή ενέργειας, υψηλή αποδοτικότητα για τη θέρμανση, την ψήξη και την παροχή ενέργειας των τοπικών κοινοτήτων. Ξεκινήσαμε επίσης και την δυνατότητα πρόσβασης στις ανανεώσιμες πηγές. Όταν τα πετυχαίνουμε όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε ένα σωστό συνδυασμό ενεργειακό, να μειώσουμε την εκπομπή διοξιδίου αντιμετωπίζουμε τα θέματα της προσαρμογής των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Το πετύχαμε από κοινού αυτό και είμαι ενθουσιασμένος θα έλεγα. Πετύχαμε επίσης να βρούμε λύσεις και σε επίπεδο δημιουργίας τοπικών θέσεων απασχόλησης, όχι μόνο την εμφάνιση των υποανάπλαση περιοχών, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μείωση της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα στις ε, εσωτερικές περιοχές των πόλεων, μείωση σχεδόν στο 40% στο εσωτερικό των περιοχών αυτών των πόλεων και μείωση επίσης και επιβεβαιώνεται και από τις δικές σας παρεμβάσεις μια σημαντική μείωση του κόστους της ενέργειας, του λογαριασμού. Ας Αυτό έχει δύο επιπτώσεις θετικές. Η μία αφορά την εξοικονόμηση χρημάτων και από την άλλη τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι στόχος και των πολύ γνωστών στόχων περιλαμβάνεται συγγνώμη στους πολύ γνωστούς στόχους της πολιτικής για την Ευρώπη του 2020. Οι πολίτες όχι μόνο θα πληρώνουν λιγότερα, αλλά θα δουν ότι η Ευρώπη κάτι πετυχαίνει για την καθημερινότητά τους. Και υπάρχουν κοινωνικά ωφέλη μέσω της δημιουργίας των θέσεων απασχόλησης οι οποίες θα δημιουργηθούν. Και υπάρχει και η οριζόντια επίπτωση στην τοπική οικονομία. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μιλάμε για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν μιλάμε για πολυεθνικές οι οποίες προσπαθούν να τοποθετούσουν ε, τα, ε, τις δυνατότητες που έχουν τις οικονομικές για να εξυπηρετήσουν τις μικρομεσαίες. Αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε στο μέλλον είναι πρώτον να υπάρξουν εθνικές στρατηγικές για να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως η κατοικία, η ανάπτυξη των πόλεων, η ανάπτυξη της υπαίθρου και οι ενεργειακές πολιτικές. Αν δεν υπάρξουν αυτές οι εθνικές πολιτικές εμείς μπορεί να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά μόνο σε πάρα πολύ μικρή κλίμακα και με μάλλον χαοτικό τρόπο. Δεύτερο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να λάβουμε υπόψη μας ότι ε, με τα χαρακτηριστικά των κρατών μελών και τις διαφορές τους, το 80% της συνοχής πηγαίνει στο Περιφερειακό Ταμείο, αλλά τα υπόλοιπα θα πρέπει να καλυφθούν από το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο και αν είναι απαραίτητο για αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο, για αυτούς που θίγονται από τη φτώχεια, να χρησιμοποιηθεί και το κοινωνικό ταμείο για να καλυφθούν οι υπόλοιπες ανάγκες και να βελτιωθούν οι συνθήκες κατοικίας τους. Δεν έχω άλλες παρατηρήσεις, σύντομες παρατηρήσεις, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και ευχαριστώ τους ερευνητές διότι πράγματι δείχνουν ποια είναι τα ωφέλη της, της ε, κοινωνικής μας πολιτικής στο συγκεκριμένο τομέα. Κοιτάξτε κυρία Μανέσκου, αν, αν μιλήσετε πολλή ώρα δεν θα υπάρχει διαμηνία για την παρέμβαση του Νίκου. Ε. Θα είμαι σύντομη. Καταρχάς να συγχαρώ τους δύο ερευνητές. Δείχνουν ότι πράγματι το θέμα αυτό είναι ευρωπαϊκό θέμα είναι θέμα το οποίο και εμείς τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να προωθήσουμε με διαφορετικά ποσοστά επιτυχίας. Πρόκειται για ευρωπαϊκό θέμα και χαίρομαι που το ανέφερε και ο κύριος Τσέλερ. Έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Οι προκλήσεις αυτές δεν αφορούν μόνο τα παλιά κρατημέλη αλλά και τα νέα κρατημέλη, αντίθετα μάλλον. τα νέα κράτη-μέλη είναι πραγματικά σε μειονεκτική θέση, πιέζουν συνεχώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να βοηθηθούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της κοινωνικής κατοικίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί μιλάμε για κατοικίες οι οποίες έχουν οικοδομηθεί στη δεκαετία του 60 και υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα με το κόστος της θέρμανσης, του ηλεκτρισμού, των επιπέδων ζωής, της ποιότητας ζωής κτλ. και οι επιπτώσεις των παρεμβάσεών μας και η επιτυχία τους στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι αλήθεια ότι επίσης κατά τη διάρκεια ε, της επομένης περίοδου στο εσωτερικό του Περιφερειακού Ταμείου έχουμε πολλές δράσεις για την ανάπλαση των κέντρων των πόλεων μέσω των ολοκληρωμένων ε, ε, εδαφικών επενδύσεων. Απαιτείται να υπάρχουν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Έχουμε κανόνες ξεκάθαρους, έχουμε το Ταμείο Συνοχής, το οποίο για πρώτη φορά θα είναι ανοιχτό σε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα και θα συνεισφέρει άμεσα στα προβλήματα της κατοικίας. Έχουμε τα χρηματοδοτικά μέσα αυστηρά του ταμείου μας, του Περιφερειακού Ταμείου και όχι μόνο με τα μέσα αυτά, όχι μόνο με το Ταμείο Συνοχής, μπορούμε παρόλα αυτά να ασχοληθούμε και με τις δυνατότητες που παρέχει η Τζέσικα και άλλα μέσα. Έτσι ώστε να καταστούμε πιο αποδοτικοί ενεργειακά και να μην παραμείνουμε σε ένα θεωρητικό επίπεδο αλλά να εφαρμόσουμε σωστά αυτή την πολιτική, μια σημαντική πολιτική και τα επόμενα χρόνια με τις δημοσιονομικές πιέσεις που υπάρχουν αυτά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα πράγματι τα έχουμε πολύ ανάγκη ε, και ένα παράδειγμα είναι η Τζέσικα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για μια ακόμη φορά που καταστήσατε αυτή την προσπάθεια εφικτή. Νίκο παρακαλώ σύντομα. Θέλω να επισημάνω μερικά σημεία τα οποία αναφέρατε. Yes, I like to, to repeat remarks. Ε, αυτοί που χρειάζονται περισσότερα, περισσότερο αυτά τα προγράμματα είναι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αλλά είναι και αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν τις αιτήσει για τα προγράμματα. Εάν εξασφαλίσουν, αν ας πούμε ότι κάνουν τις αιτήσει, έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και αν εξασφαλίσουν συγχρηματοδότηση, τα επιτόκια είναι πάρα πολύ ψηλά. Επομένω, αυτοί που χρειάζονται παρόμοιε παρεμβάσει, είτε μονομένα είτε σε γειτονιέ ολόκληρε, έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία. Εάν υπάρχουν ε, υποστηρικτικά σχήματα από την αυτοδιοίκηση, μπορούν να αντιμετωπιστούν να περιοριστούν τα προβλήματα. Αν όμω και η αυτοδιοίκηση δεν είναι σε θέση να βοηθήσει, να στηρίξει αυτέ τι προσπάθειε, τότε έχουμε πλήρη αδυναμία να ε, κατευθυνθούν αυτά τα προγράμματα σε αυτούς που τα χρειάζονται. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που το βλέπουμε σήμερα που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν λογαριασμούς, ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές και τα χτίρια είναι πολύ παλιά και δεν αρκεί όπως υπόθηκε μόνο ενεργειακή παρέμβαση αλλά χρειάζεται μια συνολική ανακαίνιση των κατοικιών αυτών. Και τέλος υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που ήδη εντοπίστηκε και από άλλους συναδέλφους. Οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται ότι αν ανακαινιστούν οι γειτονιέ του, θα φύγουν από τι γειτονιέ. Και πράγματι αυτό συμβαίνει πολλέ φορέ γιατί ανεβαίνει το κόστο των χτιριών και των υποδομών, άρα στο τέλο νιώθουν εχθρικοί σε προσπάθειε ανακαίνιση. I understand there was no criticism of Κατάλαβα ότι δεν έγινε, ε, διατυπώθηκαν επικρίσεις κατά των ε, ε, μελετών σας, αλλά θέλετε να πάρετε το λόγο παρόλα αυτά. Σύντομα, ευχαριστώ πολύ για τα θετικά σας σχόλια. Πρώτον, η κυρία Σάντσες μίλησε για 20 δις. Εμείς υπολογίσαμε 1,5 δις για τη στέγαση είναι λοιπόν πολύ μικρότερα τα ποσά, αλλά παρόλα αυτά ε, όχι ευκαταφρόνητα. Ο κύριος Όλμπριχτ ρώτησε ποιες θα είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις. Δεν ξέρουμε, γιατί δεν τις έχουμε μετρήσει ακριβώς. Πρώτον, να ενθαρρύνουμε ε, τους ε, νομοθέτες να είναι πολύ συγκεκριμένοι στο πώς θα καθορίσουν τους ε, δείκτες Και το τρίτο που είπε ο κύριος Τσέλερ, ναι, τα κάναμε όλα αυτά, αλλά δεν θα μειωθεί ο λογαριασμό σα γιατί έχουν εκτοξευθεί οι τιμέ τη ενέργεια. Ακριβώ. Πρέπει να του πούμε ότι αν δεν είχαν γίνει αυτές οι επενδύσει, τότε ο λογαριασμό του θα ανέβαινε ακόμη πιο πολύ. Αυτό πρέπει να του υποθεί. Καταλαβαίνουμε βέβαια την απογοήτευση των ε, κατοίκων που διαπιστώνουν ότι δεν μειώνεται ο λογαριασμός τους. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή για την ε, ε, περαιτέρω διανομή αυτής της μελέτης. Η κυρία ε, Βίντσοβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε και αποδεικνύεται πάντοτε τελικά ότι είναι πολύ ευρύτερο το πλαίσιο και πολύ, πιο πολύπλοκο το όλο θέμα. Αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω δύο-τρία πράγματα σε ό,τι αφορά την τομική προσέγγιση για το μέλλον. Έχουμε τώρα κάποιες, ε, ε, κάποια στοιχεία για το παρελθόν, αλλά να πάμε στο μέλλον. Τώρα για τα 20 δις, δεν ξέρω ακριβώς πώς έχει υπολογισμό, ε, το 5% από το ΕΤΠΑ, ίσως είναι λίγο λιγότερο. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή τα ποσά. Σε ό,τι αφορά όμως την τομιακή προσέγγιση, καθώς και το ζήτημα της επικουρικότητας για ε, χαμηλότερο επίπεδο. Η στέγαση από την πλευρά της πολιτικής συνοχής πρέπει να πούμε ότι είναι ένα εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε άλλα θέματα. Δεν είναι δηλαδή η στέγαση ε, ο αυτός Απλά ε, είναι το μέσο για την επιτεύξη άλλων στόχων, ένα εκ των οποίων είναι η ενεργειακή απόδοση και αυτό γιατί έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είναι 40% των εκπομπών του ε, διοξιδίου του άνθρακα ε, που έχουν σχέση με την ενεργειακή απόδοση. Ένας αυτός ο στόχος. Δεύτερος στόχος, κοινωνική ένταξη. Θέλουμε λοιπόν αυτού τους δύο στόχους να τους πετύχουμε και να τους συνδυάσουμε. Καταλαβαίνω και συμφωνώ. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη στέγαση μία φορά για την κοινωνική ένταξη και την επόμενη φορά για την ενεργική απόσπαση. Πρέπει να έχουμε μια ε, συντονισμένη προσέγγιση όταν λοιπόν έχουμε ολοκληρωμένε δράσει για την αστική ανάπτυξη, μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Πολλέ φορέ ακούσαμε να γίνεται λόγο για στρατηγική προσέγγιση. Εδώ πράγματι η αστική διάσταση για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, αυτό το 5%. Θέλουμε να είναι τουλάχιστον 5% και να σχετίζεται με μια στρατηγική προσέγγιση. Να έχουμε δηλαδή κάλυψη και των 5 πτυχών. Άρα, η στέγαση, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι πολύ απλό θέμα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με συντονισμένο τρόπο, με μια συντονισμένη προσέγγιση, έτσι ώστε να φέρει τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι πώς το προσεγγίζουμε σε συνεργασία με το τοπικό επίπεδο, να δώσουμε δυνατότητες στην τοπική κοινότητα. Πολύπλοκα και δυσεφάρμοστα όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον από ρυθμιστική πλευρά πιστεύω ότι πλέον ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά και μέσω της άσκησης ε, του προγραμματισμού για φέτος εξασφαλίσαμε να αντιμετωπίσουν σωστά αυτά τα προβλήματα ε, σε αυτό το πλαίσιο. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, είμαστε όμως ανοιχτοί και μπορούμε να συστήσουμε ενδεχομένω μελλοντικά ε, και πάλι αυτό το θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, ήταν πολύ το feedback, να ευχαριστήσω βέβαια και τους ερευνητές που μας έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να ευχαριστήσουμε τους εμπειρογνώμονες, ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λίγη λοιπόν ε, σήμερα η συνάντησή μας, 10 και 11 ε, Ιουλίου θα συνεδριάσουμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ. Λίγη τη συνεδρίαση.